Euh, Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Έχουμε μια ακρόαση κοινή σήμερα, οι δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές ΚΡΙΜ και ΛΥΜΠΕ για την προσαρμογή των δομών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ε, στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και του ξεπλήματος χρήματος. Λοιπόν, στα πλαίσια της πρώτης συζήτηση, σε αυτή την ε, κοινή μεικτή ακρόαση, θέλουμε να ενισχύσουμε τις βάσεις του ποινικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, ποινική δικαιοσύνης και γι' αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε με την, ε, με την κυρία Ρέντινγκ, που είναι η επίτροπος υπεύθυνη για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίασή μας. Προτείνω να οργανώσουμε τη συζήτησή μας ως εξής. Ο κύριος Αγγιλέρ θα έρθει σε λίγα λεφτά. Θα γίνει μια παρουσίαση 30 λεπτών από την κυρία Ρέντινγκ και συνεχεία θα γίνει ένας πρώτος γύρος ερωτήσεων από τους ευρωβουλευτές που θα έχουν ζητήσει το λόγο. Θα δοθεί προτεραιότητα στον εισηγητή, στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και των δύο επιτροπών, και Λίμπε και Κρίμ δηλαδή. Και θα ήθελα ο καθένας να περιοριστεί σε Δύο λεπτά παρακαλώ. Και η κυρία Ρέντινγκ θα έχει μία ώρα για να απαντήσει. Και αν έχουμε αρκετό χρόνο, θα ακούσουμε και δεύτερο γύρο ερωτήσεων από τους ευρωβουλευτές. Θα απαντήσει βεβαίω η κυρία Ρέντινγκ και συνεχεία θα συνεχίσουμε το δεύτερο και τρίτο πάνελ. Κυρία Πίτροπ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, όλοι γνωρίζετε επειδή δουλεύετε επ' αυτού ότι προκύπτει ένας νέος ποινικό ορίζοντας στην Ευρώπη. Το οργανωμένο έγκλημα αλλάζει, γίνεται πιο ποικιλόμορφο τις μεθόδους του, στο πώς οργανώνεται και στις επιπτώσεις του στην κοινωνία. Η πρόσφατη αξιολόγηση της Europol για την απειλή από το οργανωμένο έγκλημα επιβεβαιώνει ότι σε πολλά κράτη-μέλη, σε πολλές δικαιοδοσίες και σε πολλούς τομείς έχουμε τέτοια φαινόμενα. Προσπαθούμε να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα εδώ και πολλά χρόνια με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και το ξέπλυμα του χρήματο, αλλά για να είναι αποτελεσματικό ο αγώνα, χρειαζόμαστε μια πολύ σχηδή προσέγγιση. Και το ποινικό δίκαιο εδώ μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει να προστατεύει τις κοινέ αξίες, τα κοινά αγαθά μας και θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα σοβαρά ποινικά δικήματα που παραβιάζουν αυτές τις αξίες προβλέπονται, διερευνώνται, διώκονται και όχι μόνο στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για να καταπολεμήσουμε το σοβαρό οικονομικό έγκλημα με διασυνοριακή διάσταση, αυτό ε, είναι ε, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρεται στην α, ε, Συνθήκη της Λισαβόνας. Όμως, εκατομμύρια ευρώ μπαίνουν σε λάθος α, τσέπες εξαιτίας εγκληματικών δραστηριοτήτων. Το έγκλημα γίνεται πιο περίπλοκο. Συχνά οι, διαστα... διαστάσεις του είναι διασυνοριακές, επομένως είναι δικαιοδοσία περισσότερων κρατών μελών. Μερικές φορές επηρεάζονται και τα κρατημέλη και οι πολίτες και οι εταιρείε. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται δράση και η Κομισιόν έχει κάνει ορισμένα πράγματα. Έχουμε την οδηγία κατά της απάτης καταρχάς. Έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε την απάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μία θέλουμε να ενισχύσουμε το νομικό πλαίσιο, να το ενοποιήσουμε και από την άλλη να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στα κείμενα που σκοπό έχουν να προστατεύσουν τα χρήματα φορολογουμένων από τη διαφθορά και την κατάχρηση. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Γιατί ξέρετε ότι πάνω από 90% του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης το διαχειρίζονται οι εθνικές αρχές. Και δεν είναι τυχαίο που υπάρχουν απάτες σε, εθνικά, σε εθνικό επίπεδο, όπου η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετική από κράτος σε κράτος. Επομένως, αυτός ο κατακαιρματισμός πρέπει να ξεπεραστεί και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά χρήματα που επενδύονται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ε, αντιμετωπίζονται έχουν την ίδια αξία παντού ε, και καταπολεμάται η απάτη με τον ίδιο τρόπο. Εγώ έχω γράψει τον όρο «Μηδενική ανοχή» στη σημαία μου. Τον Ιούνιο του 2012 πρότεινα μια οδηγία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου και το καταφέραμε αυτό χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας, αυτό το κείμενο δηλαδή, όπου υπάρχει μια βάση για το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο που μπορεί να καταπολεμήσει τις παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, πλήρη συναπόφαση για το Κοινοβούλιο και επομένω είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να αρχίσει να εργάζεται επί του θέματος αυτού, ούτω ώστε να χρησιμοποιήσουμε πλήρω τη συνθήκη και τα πλεονεκτήματα που μας δίνει. Έχουν περάσει πάνω από 6 μήνες τώρα, από τη στιγμή που κατατέθηκε η πρόταση ενώπιον του Κοινοβουλίου και καλό θα ήταν το Κοινοβούλιο να προχωρήσει και να αναλύσει αυτή την πρόταση. Η συνθήκη προβλέπει μια νομική βάση για μέτρα ad hoc, διοικητικής και ποινική φύσεως, και τα δύο δηλαδή, και επιτρέπει κατά συνέπεια την ομοιόμορφη προστασία σε όλα τα κράτη-μέλη δηλαδή. Αυτό που γράφει αυτή η πρόταση δηλαδή είναι το εξή. Καταρχάς, εισάγουμε κοινού ορισμού για τα παραπτώματα δικήματα κατά του κοινοτικού προπολογισμού, του νοσιακού προπολογισμού. Επομένω, θα έχουμε κοινή προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο των οικονομικών συμφερόντων. Ένα παράδειγμα, η κατάχρηση των διαδικασιών των προμηθειών με σκοπό τη διάπραξη απάτης αυτό προβλέπεται στην νομοθεσία κάποιων κρατών μελών, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη δεν προβλέπεται αυτό. Επομένω, οι κοινοί ορισμοί θα πετύχουν μια, ένα ενίο επίπεδο προστασία και θα κλείσουν τα παραθυράκια τα οποία χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή οι εγκληματίες, γιατί οι εγκληματίες γνωρίζουν το δίκαιο και φυσικά επιλέγουν τον τόπο όπου δεν τους παρεμποδίζει κανείς ε, για τη διάπραξη των εγκλημάτων τους. Μια άλλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αφορά τις ε, ελάχιστες κυρώσεις. Κάποια κράτη-μέλη έχουν τέτοιες ελάχιστες κυρώσεις, ενώ άλλα όχι. Και αυτό οδηγεί σε θέματα διατησίας. Όταν ε, βρίσκουν οι εγκληματικές οργανώσεις ε, ασφαλείς τόπους, παραδείσους για να προβούν στι δραστηριότητε τους. Εγώ προτείνω ελάχιστη κύρωση, έξι μήνες φυλάκιση για τα σοβαρά δικήματα. Όταν υπάρχει βέβαια ε, σοβαρότατη ζημία στο, κατά του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή πολύ υψηλά κέρδη ε, των δραστών. Αυτό θα είναι ένα αντικίνητρο και ελπίζουμε θα παρεμποδίσει τους απαταιώνες και επιπλέον τα κράτη-μέλη θα είναι υποχρεωμένα να έχουν ε, κοινού κανόνες για τα όρια παραγραφής στις ποινικέ δίκες. Δηλαδή την περίοδο μετά την οποία δεν μπορείς πια να διώξεις κάποιον. Γιατί πολλοί εγκληματίε χρησιμοποιούν την ε, τακτική της παρακόλλησης, αφήνουν το ρολόι να τρέχει, ούτως ώστε να διαφύγουν του νόμου. Θέλουμε να σταματήσει αυτό. Αυτή η οδηγία κατά τη απάτηση είναι μια πρώτη σημαντική πράξη για πιο αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο συζητείται στο Συμβούλιο από το περασμένο καλοκαίρι και προσβλέπω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αρχίσει τις εργασίες του επ' αυτού του κειμένου. Και κάνω πραγματικά έκκληση εδώ στην Επιτροπή σας, ο εισηγητής να οριστεί το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αρχίσει η δουλειά από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι εγκληματίε δεν έχουν κανένα σεβασμό, πρέπει να σα πω, για το ποιος, ποιο θεσμικό όργανο ε, έχει την αρμοδιότητα εδώ και ποιο εκεί. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τη θεσμική διάσταση ως εγγυητή για την προαγωγή ε, ευρωπαϊκής πολιτικής. Θα θυμάστε ότι μίλησα στην ακρόασή μου για αυτό το θέμα και θα το ξαναβάλω επιτάπητος τους επόμενους μήνες. Επίσης, ε, και τι σημαίνει αυτό, σημαίνει το, Ευρωπαϊκό, το γραφείο του Ευρωπαίου, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για να έχουμε ε, επιτυχή δίωξη των εγκληματιών κατά ε, των των εγκληματιών κατά των οικονομικών σπρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θα πρέπει να, έχουμε, ε, να μην έχουμε το λεγόμενο ελβετικό τυρί. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε μειώμενη προστασία. Γιατί η προστασία παίζει πάρα πολύ. Από το 19% προστασία στο, ως το 90%. Τεράστια διαφορά από κράτος σε κράτος λοιπόν. Ο προπολογισμό όμως είναι κοινό. Ε, ευρωπαϊκοί φορείς όπως η Europol ή η Eurojust μπορούν να βοηθήσουν, μπορεί να συντονίσουν τις διασυνοριακέ έρευνε και διώξεις. Αλλά δεν μπορούν ούτε να εκκινήσουν, να δρομολογήσουν δηλαδή, ούτε να κατευθύνουν έρευνες. Επομένως αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, το άρθρο 86 όλους ιδιαίτερος, που προβλέπει την δημιουργία ενός, ενός γραφείου Ευρωπαϊκής Αγγελίας, ε, υπεύθυνου για την έρευνα, δίωξη και εκδίκαση των απαταιώνων που πλήττουν τον ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό. Έχουμε προχωρήσει τις διαβουλεύσεις και τις προτάσεις και η πρόταση θα κατευθύνεται στο καλοκαίρι. Θα έχει μια σαφή εστίαση στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ποια θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Η συνθήκη λέει ότι το γραφείο αυτό του Ευρωπαίου Εισαγγελέου θα δημιουργηθεί από τη Eurojust. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε στενές σχέσεις μεταξύ του γραφείου αυτού και της Eurojust και θα πρέπει να υπάρχουν ε, λειτουργικές, ε, επιχειρησιακές και διοικητικές ε, επαφές. Θα πρέπει να έχουν αποκεντρωμένο, ολοκληρωμένο σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, αυτό το γραφείο θα είναι ένα ευρωπαϊκό γραφείο, αποκεντρωμένο, που σημαίνει ότι αυτό το γραφείο επιχειρησιακά θα ανήκει στα κράτη-μέλη και θα ερευνά άμεσα, θα διώκει και θα εκδικάζει σε, όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα δικήματα κατά των ευρωπαϊκών συμφερόντων μαζί με τις ε, εθνικές δικαστικές αρχές και τις ε, διοκτικές αρχές. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να οργανώσουμε τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των εθνικών αρχών, ούτως ώστε να μην έχουμε επικαλύψεις των εργασιών. Το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα έχει αυτόνομες ε, εξουσίες έρευνας και δίωξης και θα πρέπει να έχουμε ασφαλιστικές δικλείδες για την ανεξαρτησία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ανεξαρτησία και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και από τις εθνικές αρχές. Και αυτή η ανεξαρτησία θα αυξήσει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την νομιμότητά της. Παράλληλα, θα λογοδοτεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν λόγο ε, στο, στις επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Η επιχειρησιακή επίσης αυτονομία θα πρέπει να εξασφαλιστεί, ενώ όλες οι έρευνες θα υπόκεινται σε αυστηρό δικαστικό έλεγχο. Πολύ σημαντικό επίσης, η Ευρωπαϊκή Αγγελία θα πρέπει να έχει μικρό προσωπικό, ε, να μην είναι δαπανηρή. Θα πρέπει η σχέση κοστος ωφέλους να είναι πολύ επωφελής. Θα πρέπει να υπάρξουν οικονομίες κλίμακας. Θα πρέπει να επιτεθούμε στην απάτη, αλλά με χαμηλό κόστος. Δηλαδή, θα έχει προσθέμενη αξία, θα φέρει αλλαγές στον κύκλο της εφαρμογής του νόμου, της ανείχνευσης, της δίωξης, της δίκης. Και αυτός ο κύκλος μέχρι στιγμής ήταν αδύναμος κατακαιρματισμένος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα εξασφαλίσει την, θα εξασφαλίσει την ε, ενότητα ε, και την αποτελεσματικότητα σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, κάτι που συνδέεται με αυτό. Και σας έχω ήδη αναφέρει το άρθρο της ε, συνθήκης, το σχετικό. Συνδέεται λοιπόν η συνεργα... με αυτό το θέμα η συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Αγγελία. Η πρόταση για τη δημιουργία ενός τέτοιου γραφείου θα συνοδεύεται από μια πρόταση για τη μεταρρύθμιση της Eurojust. Είναι το τρίτο ορόσημο της ολοκληρωμένης μας προσέγγισης, η προτινόμενη μεταρρύθμιση της Eurojust που θα αντιμετωπίζει και τα θεσμικά και τα πρακτικά θέματα και τις σχέσεις μεταξύ Eurojust και Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Από τη στιγμή της γέννησης της, η Eurojust ε, γνώρισε σημαντικές εξέλιξεις και αλλαγές. Ξεκίνησε το 2000, σαν ένα άτυπος, ας πούμε, μια άτυπη συνάντηση των εισαγγελέων. Αλλά στην πραγματικότητα έγινε πραγματικός, σύν το χρόνο δηλαδή, έγινε πραγματικός ε, παίχτης, φορέας στην, ε, σε θέματα ποινική δικαιοσύνη. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε από την εικόνα τη Eurojust. τελευταία χρόνια η Eurojust ε, έπαιξε ρόλο για το συντονισμό διασυνοριακών ε, ερευνών σοβαρών αδικημάτων και για το, τη διαφθορά και για το οργανωμένο έγκλημα και για το ξέπλυμα του χρήματος. Το 2011 το Eurojust ε, διοργάνωσε 204 συναντήσεις συντονιστικές και διοργάνωσε 33 κοινέ ε, ερευνητικέ επιτροπέ. Μην ξεχνάμε όμω ότι μπορούμε να επιτύχουμε περαιτέρω πρόοδο, γίνεται και είναι και επιθυμητό και πιστεύω ότι μπορούμε να ετοιμάσουμε τη Eurojust για τη νέα ε, δεκαετία δικαστική συνεργασία, να εξυγχρονίσουμε το δικαστικό τη πλαίσιο, να απλουστεύσουμε τη λειτουργία τη και τη δομή τη, να την κάνουμε πιο διαφανή και πιο πιο ελεγχόμενη, γιατί αυτό το απαιτεί και η συνθήκη της Λισαβόνας και ξέρετε ότι η Eurojust δημιουργήθηκε ως τρίτος πυλώνας. Είχε δημιουργηθεί μάλλον ως τρίτος πυλώνας πριν υπάρξει η συνθήκη της Λισαβόνας. Θα πρέπει τώρα αυτό το όργανο να γίνει πιο δημοκρατικό, πιο διαφανές, όπως το προβλέπει η Λισαβόνα και να δώσουμε ε, σαφή ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust. Επομένως, είναι ένα θέμα που επανέρχεται συνέχεια και μπαίνει σε όλες τις νέες προτάσεις ε, που υποβάλλονται. Και η Eurojust θα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική φυσικά. Αυτό σημαίνει μείωση του διοικητικού άχθους των ε, κρατών μελών και να τους επιτρέψουμε να ασχοληθούν πραγματικά με τα βασικά τους ε, καθήκοντα που είναι η καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος. Επομένως, η μεταρρύθμιση θα εισαγάγει ένα μηχανισμό για να διαχωρίσουμε καλύτερα μεταξύ του επιχειρησιακού κομματιού και του διοικητικού κομματιού. Θα δούμε το ρόλο και την ευθύνη όλων των φορέων και τον ποιες είναι οι ευθύνες επίσης των εθνικών μελών ε, του κολεγίου. Θα δούμε το νομικό καθεστώς, θα έχουμε ένα νέο κανονισμό, ο οποίος θα είναι εφαρμοστέως απευθείας όλα τα κράτη-μέλη και με αυτόν τον τρόπο οι δύσκολε νομικέ δομέ ε, που έχουμε σήμερα θα ξεπεραστούν. Χρειαζόμαστε μια ενοποιημένη, ολοκληρωμένη προσέγγιση για να καταπολεμήσουμε την ε, ευρωπαϊκή απάτη. Το ξέρετε. Προσπαθώ να το πετύχω. Ε, Υποβάλλοντα, μια και είμαι επίτροπο ε, για θέματα δικαιοσύνη και με τη νέα μου αρμοδιότητα για το ποινικό δίκαιο, αυτές τις προτάσεις που σας παρουσίασα και άλλες όμως. Και πιστεύω ότι αυτό το πακέτο θα δώσει μια νέα ορμή στον αγώνα κατά της, του εγκλήματος και της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε την Επίτροπο. Ε, κύριε Αγγιλάρ, θέλετε να πείτε δύο λόγια. Παρακολούθησα την εισήγηση αυτή για τις προοπτικές αυτές διασύνδεσης των προσπαθειών που ε, γνωρίζει η Europol και η Eurojust, έτσι ώστε να ενώσουμε αυτές τις προσπάθειες για την δικαιοδοτική συνεργασία σε θέματα που άπτονται του ποινικού δικαίου. Η πρωτοβουλία αυτή σχετίζεται με τη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Εισαγγελικής Αρχής, που θα πληρεί τους όρους που έχουν αναφερθεί στο άρθρο 86 της Συνθήκης Περιλειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχουν πολλές ε, προκλήσεις ενώπιον μας και που ε, κατατροπώνουν τα κράτη-μέλη ένα προς ένα καθε αυτά. Τα βαρύνουν ιδιαίτερα. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταβάλει μια προσπάθεια για τη σύσταση μιας οδηγίας για την προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παρούσα κατάσταση δεν έχει διασαφιστεί ακόμα. Η Γιούρι, η Λίμπε και η... By Και Κοντ συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και αναμένουμε και από την ΚΟΝΤ να γνωμοδοτήσει. Εάν δεν ξεδιαλύσουμε αυτό τον μύτο και δεν ε, βγούμε από την κατάσταση ε, αυτού του αδιεξόδου, θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα πριν από τη λήξη της θητείας και αυτό θα ήταν πολύ αρνητικό μήνυμα. Νομίζω ότι οι πολίτες ε, αναμένουν συνεργασία σε θέματα δικαστικών αρμοδιοτήτων και πρέπει να δείξουμε στο Συμβουλίο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να νομοθετήσει επί της ουσίας όσον αφορά ζητήματα που άπτονται του ποινικού δικαίου και να κάνει ένα βήμα προς τα μπρος σε θέματα χρηματοοικονομικού συμφέροντος. Με βάση την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αναλυφθεί και που θα πρέπει να ολοκληρωθεί και εγώ ως εισηγητής από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να συνεργαστώ και με τις δύο επιτροπές ε, με βάση τον, το άρθρο 49 του κανονισμού και θέλουμε να καταδείξουμε στην Επιτροπή ότι οφείλουμε να συνεργαστούμε πριν από τη λήξη της θητείας, ε, συνάδελφοι, έχουμε μισή ώρα για τις ε, ερωταποκρίσεις. Η κυρία Ματιέ έχει το λόγο καταρχήν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά σας ε, βρίσκουμε εδώ ενώπιόν μας, κυρία Επίτροπε. Βλέπετε ότι το Κοινοβούλιο κάνει ό,τι μπορεί για την αντιμετώπιση της ε, διαφθοράς και των αποτελεσμάτων της. Και αυτό ιδιαίτερα έναντι τρίτων χωρών. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ανέκυψε αυτή η Ειδική Επιτροπή Κρίν στα πλαίσια της Επιτροπής ΛΥΠΕ. Συστάθηκε δηλαδή από την Επιτροπή ΛΥΠΕ και γι' αυτό βρίσκεστε εδώ ενώπιόν μας. Χαιρόμαστε για την πρόταση, την πρότασή σας οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος και ο πρόεδρος Λόπες Αγγιγιάρ μίλησε για την κατάσταση αποκλεισμού που υπάρχει, που υφίσταται τώρα και με μεγάλη χαρά θα συμμετάσχουμε στην όλη διαδικασία διασάφησης του ζητήματος. Ως προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, αναμένουμε τις προτάσεις σας. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε μία καταληκτική ημερομηνία. Πότε θα λάβουμε δηλαδή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί την αναμένουμε εδώ και καιρό. Δεν νομίζω θα καθυστερήσει άλλο με μεγάλη μας ε, χαρά και εύνοια θα την ε, δεχτούμε. Γνωρίζουμε εδώ και ένα χρόνο μετά τη σύσταση της Επιτροπής ΚΡΙΜ και ακροάσεις της Europol και της ΕΠΟΛ, επειδή ακριβώς προσήλθαν πολλοί εμπειρογνώμονες και μας εξήγησαν την κατάσταση, γνωρίζουμε και έχουμε συνειδητοποιήσει τη διάσταση αυτής της διαφθοράς ενώ πολλά κράτη-μέλη ε, δεν ξέρουν ε, τις ομάδες ε, μαφίας που λειτουργούν μέσα στα κράτη-μέλη και διασυνοριακά με γιατί αυτό το είδαμε και στην ΔΕΒ σήμερα το πρωί σε μια κοινή ακρόαση. Εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλλετε και νέες προτάσεις. Ο ρόλος μας είναι σημαντικός όπως και του Συμβουλίου. Αναμένουμε νέες προτάσεις, πιο συγκεκριμένες, και οι οποίες να μας δώσουν κατευθυντήριες γραμμές. Νιούτον Ντάν. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση ήταν η δική σας, κυρία Επίτροπε. Εγώ επειδή είμαι φιλοευρωπαϊστής, κατανοώ ότι μιλήσετε για μια νέα εικόνα που διαγράφεται. Ε, βρισκόμαστε μεσοστρατής ακόμα. Δεν ε, έχουμε παρά την εθνική αστυνομία, τις εθνικές φυλακές, τις εθνικές ανακριτικές αρχές και ούτω καθεξής. Εσείς πιστεύετε ότι θα υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και μία αρχή τύπου FBI. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την Επίτροπο για την ε, παρουσίασή της. Εδώ και ένα χρόνο είδα μία έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς μία ε, ευρωπαϊκή προσέγγιση για το ποινικό δίκαιο όπου αναφέρεται ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς το ποινικό δίκαιο και να βασιζόμαστε σε πραγματικά γεγονότα και στοιχεία για να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ουσιαστικό διασυνοριακό στοιχείο. Και ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τα, τα ασφαλή ε, λιμάνια, όπως τα ορίσατε για τους εγκληματίες. Όμως δεν υπάρχουν απτά αποδεικτικά στοιχεία εγκληματικής δραστηριότητας, crime shopping στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε αυτά αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι εγκληματίες περνάνε σε μία χώρα και δρούν σε μία χώρα όπου ε, οι κυρώσεις είναι χαμηλότερες, γιατί αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αυτό είναι ένα πολύ καλό επιχείρημα για τα κράτη-μέλη που δεν θέλουν να εναρμονίσουν το ποινικό δίκαιο. Διαφορετικά δεν μπορούμε να δράσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ευπρόσδεκτες βεβαίως είναι όλες οι πληροφορίες. Ένα άλλο στοιχείο έχει ως εξή. Στην έκθεση του Κοινοβουλίου φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν οριζόντια στοιχεία του ποινικού. Και αναφέρθηκα σε μερικά. Μιλάμε για ελάχιστες ε, κυρώσεις. Εάν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά όχι για ένα είδος εγκλήματος. Χρειαζόμαστε πιο οριζόντιες ε, συζητήσεις για να ε, δώσουμε προστιθέμενη αξία στις ευρωπαϊκές αξίες δηλαδή να μην αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα εγκλήματα, αλλά γενικότερα σε ένα ευρύ πλαίσιο παραπτωμάτων. Και μιλήσατε για την παραγραφή των εγκλημάτων. Επίσης, ένα άλλο οριζόντιο ζήτημα είναι το στάτους της παραγραφής. And also to, to agree at European level what... Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς έχει το καθεστώς της παραγραφής, ιδιαίτερα για μείζωνα εγκλήματα. Και άλλα ζητήματα θα ανακύψουν μέσα στα πλαίσια ε, της έκθεσης αυτής, δηλαδή ως προς την, ε, το κατά πόσο είναι υπόλογα ε, ποινικά τα νομικά πρόσωπα. Και ένα άλλο ζήτημα είναι ότι υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση ποινικών κυρώσεων, αλλά όχι διοικητικών. Και αυτό θέτει όλο ένα και μεγαλύτερα προβλήματα μέσα στα πλαίσια τις θέσεις σε ισχύ ενός νέου καθεστώτος για την... Ευχαριστώ κύριε Ντεγιούγκ, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο επόμενος ομιλητής παρακαλώ. η πρώτη ερώτηση είναι ακριβώς αυτή. Ε, καταρχάς χαίρομαι για αυτή την πρόταση που κάνετε για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και εγώ θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα γιατί αυτό το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και ακούγεται πολύ. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Αν υπάρχει ιδέα να προωθήσουμε ε, καταρχάς γενικούς κανόνες για θέματα διαφθοράς στην Ευρώπη, προκειμένου να αφυπνίσουμε την κοινή γνώμη πέρα από τα θεσμικά όργανα για τις επιπτώσεις της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Ειδικά σε αυτή τη φάση της οικονομικής κρίσης, ε, τι επιπτώσεις έχει λοιπόν στις επιχειρήσεις και, τον, και στις κοινωνίες μας. Κομισιόν, πριν από το 2014 θα υπάρξει ευρωπαϊκό ραντεβού, ούτως ώστε να είναι την άποψή του όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάρλερ. Μετά ο κύριος Γιακολίνο, εισηγητής μας. Και ο κύριος Μέρα. Και τελευταίος βεβαίω ο Επίτροπο. Ε, κυρία Βάιλερ, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύο σύντομε ερωτήσει έχω. Η πρώτη αφορά κάτι που η συνάδελφος Ματιέ είπε πριν. Σε όλες τις ακροάσεις μας κατά το τελευταίο έτος είχαμε την σύσταση και από Αμερικανούς και από τον ΟΣΑ και από τον ΟΗΕ από όλους τους επαΐοντες είχαμε τη σύσταση οπωσδήποτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε πιο εμβαθυμένη συνεργασία, πιο έντονη συνεργασία μέσα σε ένα ενιαίο σύστημα παράδειγμα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή κάτι τέτοιο σχετικό. Νομίζω θα ήταν και σχετικά απλό αν ξεκινούσαμε με την οικονομική εγκληματική πτυχή, το οικονομικό έγκλημα. Και το βλέπει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της οικονομικής κρίσης. Έχουμε και δυνάμεις που όλο και περισσότερο τα κράτη, πώς να το πω έτσι, τα εξαπατούν και εκμεταλλεύονται κάθε δυνατότητα να αποκομίσουν ωφέλη και νέοι εγκληματίες σε κάποια κράτη-μέλη. Όχι επειδή εκεί οι ποινέ είναι χαμηλότερες, αλλά επειδή υπάρχουν οπές, τρύπες εκεί, τουλάχιστον στο οικονομικό έγκλημα και τους προσφέρονται δυνατότητες να δράσουν εγκληματικά εις βάρος της Ένωσης. Έτσι πρέπει να δράσουμε λοιπόν και το δυνατόν γοργότερα να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία. Σε αυτό το πρώτο ερώτημα ακολουθεί το δεύτερο. Σε εμά τους Ευρωβουλευτές, άσχετα από ποια κοινοβουλευτική ομάδα προερχόμαστε, είναι σημαντικό να γίνει αυτό σε τούτην την κοινοβουλευτική μας θητεία. Ερώτηση, εσείς ε, έχετε κάτι, ο κύριος Μπαρόζο είχε κάποια επαφή με τα κράτη-μέλη μέχρι σήμερα με τους Υπουργούς Εσωτερικών, Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών ή Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας για να διακριβώσει και να δει πώς αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη αυτή την πρόταση. Έχουμε τη συνθήκη Λισαβόνας, δεν την ξέρουμε μέχρι τελευταίας λεπτομέρειες αλλά τουλάχιστον κάτι τέτοιο μπορεί να εμπεριέχεται στη συνθήκη Λισαβόνας. Υπάρχει κάτι όσον αφορά τους Υπουργούς Οικονομίας Οικονομικών, κάτι σχετικό που να μπορεί να δώσει συνέχεια σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βάιλερ κύριος Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Λοιπόν, ευχαριστώ κυρία Ρέντινγκ. Κυρία Επίτροπε, με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την νομοθετική πρόταση που θα απορρέει από το άρθρο 86 και που όπως και εσείς είπατε θα μπορούσε να είναι έτοιμη σε τρεις μήνες μέχρι το καλοκαίρι. Και όπως φαντάζομαι αυτή η πρόταση έχει προχωρήσει πολύ και έχω κάποιες, ε, κάποια θέματα που θέλω να απαντηθούν. Θέλω να ξέρω μέχρι, μέχρι πού θα επεκταθεί το άρθρο 86 για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο πέρα σε σχέση με αυτούς που υπονομεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να μου πείτε, είναι δυνατόν τελικά μέσα στο πλαίσιο του να αποφύγουμε επικαλύψεις, διπλό επικαλύψεις, διπλό έργο, Ποιο θα είναι ο ρόλο τη Όλαφ, τη υπηρεσία δίωξη του οικονομικού εγκλήματο, πού θα ενταχθεί η Όλαφ, θα συνεχίσει να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται σήμερα ω όργανο ή θα έχει κάποια ανεξαρτησία ή τι θα γίνει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπω γνωρίζετε, ανεπίσημα κατά κάποιο τρόπο στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε και το σχετικό σχέδιο για το, την πρόταση για τον κανονισμό για την Ευρωπόλ καθώς επίσης και για την εισαγγελία, τον Ευρωπαίο εισαγγελέα. Σύμφωνα με το άρθρο 86 θα υπάρχει μια τέτοια συνάρτηση μέσα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Eurojust. Θα έπρεπε πάλι εδώ να λάβουμε υπόψη και ένα κεφάλαιο στο νέο κανονισμό για την Ευρωπόλ που θα συμπεριλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Ευρωπόλ μέσα στο πλαίσιο αυτής της νέας διαμόρφωσης του άρθρου 86. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ κύριε Ντίας μέρα και τώρα ο κύριος Γιακολίνο, εισηγητής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Άκουσα το δεύτερο τμήμα της παρέμβασης της κυρίας ε, Ρέντι. Υπάρχουν 60 χώρες που θεωρούνται σήμερα ε, φορολογική παράδειση. Και στην Ευρώπη υπάρχουν 3.600 ε, εγκληματικές οργανώσεις. Και το 2% του ΑΕΠ, το 2 με 5% του ΑΕΠ ε, είναι χρήμα που ξεπλένεται. Ε, τρομακτικά είναι αυτά τα νούμερα. Ένας συνάδελφος πριν από λίγο μίλησε για την ανάγκη να ομογενοποιήσουμε την ευρωπαϊκή προσέγγιση, την ευρωπαϊκή στάση απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα. Στην εισήγησή μας εμείς ε, μιλάμε για το ότι προβλέπουν λίγα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν τις μαφίες. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να προβλέψουμε σε όλα τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να εκτελούμε τις ε, δικαστικές αποφάσεις. Θα ήθελα να ακούσω για αυτό το σημείο την Επίτροπο και επίσης θα ήθελα να την ακούσω για το θέμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Είναι λογικό το αίτημα να καταλάβουμε τι σχέση θα έχει η νέα εισαγγελική αρχή με τη Eurojust. Τι ρόλο θα έχει η Eurojust, τι ρόλο θα έχει η OLAF. Πιστεύουμε ότι μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να είναι γρήγορη, ευκίνητη. Ε, θέλουμε έναν Ευρωπαίο εισαγγελέα, ο οποίος ε, θα συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές. Θα θέλαμε λοιπόν να μας δώσετε κάποια στοιχεία για αυτά τα ερωτήματα. Θεωρούμε ότι η πρότασή σας... Ελπίζουμε μάλλον η πρότασή σας να φτάσει στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Και τώρα Ακόμα μια ερώτηση προς την Επίτροπο. Κυρία Ρέντινγκ, αν μου επιτρέπετε και από πλευρά μου μια ερώτηση. Ευχαριστώ. Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει την πρώτη της έκθεση για τη διαφθορά στα κράτη-μέλη. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για αυτή την έκθεση τι στοιχεία θα χρησιμοποιήσετε, ποιους δείχτες θα χρησιμοποιήσετε για να μετρήσετε τη διαφθορά, ας πούμε. Και έπειτα, ε, μιλάμε για τη διαφθορά, το ξέπλυμα του χρήματος, φαινόμενα που υπάρχουν περισσότερο στην Ανατολική Ευρώπη, λέγεται. Επίσης, κύριε Επίτροπε, είπατε ότι η κατάσταση στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ήταν κρίσιμη τη στιγμή που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσατε να μας πείτε για αυτό το πρόβλημα, για αυτό το θέμα, δύο λόγια παραπάνω. Η Επίτροπος. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω αυτά τα σημαντικά ερωτήματα, σύντομα και περιεκτικά. Ο πρόεδρος Λόπες Αγγιλάρ Κύριε Αγγιλάρ, συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν να εξομαλύνει τις εσωτερικές του διαφορές, ούτως ώστε να μπορέσει να διορίσει έναν εισηγητή για την πρόταση οδηγίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου, που έχω ήδη καταθέσει τον Ιούλιο του 2012. Ε, νομίζω ήρθε η ώρα το Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με το θέμα αυτό και να επιλύσει τα εσωτερικά του προβλήματα και διαφορές. Κυρία Ματιού, ε, μιλήσατε για την οδηγία για το ξέπλυμα του χρήματος. Είναι ένα μοθέτημα που ο συνάδελφός μου, ο Μισελ Μπαγνιέ, υπέβαλε Υπάρχουν δύο τμήματα στο πακέτο. Μία οδηγία για την πρόληψη του ξεπλήματος χρήματος και της χρηματοδότησης της χρομοκρατίας και ένα κανονισμό για την πληροφορίες, τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις, ε, τα εμβάσματα ε, των χρημάτων, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε τα ανιχνευσιμότητα των χρημάτων. Κάτι που εν μέρη απαντάει και στο ερώτημα του κυρίου Ιακολίνο. Η πρόταση που υπέβαλα εγώ αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Του προϋπολογισμού μας δηλαδή, του, ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Υπάρχει αυτή η πρόταση και καλό θα ήταν το Κοινοβούλιο να εργαστεί το συντομότερο δυνατόν επί της πρότασης αυτής. Πολλοί συνάδελφοι, πολλοί ευρωβουλευτέ με ρώτησαν πότε θα δημιουργηθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ και καιρό σχολιόμαστε. Πολύ έντονα με το θέμα αυτό. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι δεν είναι εύκολο αυτό το θέμα. Καταλαβαίνετε τι συνέπειες έχει στην ποινική δικαιοσύνη. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει για τις ε, ερευνητικές ε, αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων το να δημιουργηθεί ένα νέο φορέα. Επομένω, πρέπει να σκεφτούμε όλε τι λεπτομέρειε, όλα τα στοιχεία που αφορούν τη δημιουργία μια τέτοια αρχή. Θα είναι ένα πολύ σοβαρό νομοθέτημα αυτό. Επίσης, το άρθρο 86 της συνθήκης που προβλέπει αυτή τη δημιουργία της εισαγγελικής αρχής λέει ότι αυτό το γραφείο θα πρέπει να δημιουργηθεί για την καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Φυσικά το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του και το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει απόφαση ομόφωνα γι' αυτό. Αν αυτό δεν γίνει, αν δεν δώσει το Κοινοβούλιο τη σύμφωνη, όχι, δεν μιλάω για τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου, αλλά αν δεν υπάρξει ομοφωνία στο Συμβούλιο, τότε αυτόματα θα υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία ε, κατελάχιστον εννέα κρατών μελών, ούτω ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο, αυτό το νέο θεσμικό όργανο. Δεν πρέπει να υπάρξει ε, επιπλέον έγκριση. Επομένως, είναι ασύνηθης αυτός ο τρόπος ε, λήψης των αποφάσεων και προβλέπεται να ξεπεράσουμε τα όσα προβλέπει το άρθρο 86 που μιλάει για την καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Αυτή η υπέρβαση είναι δυνατή σε σχέση με το άρθρο 86 αλλά είμαστε στη φάση της ομοφωνίας του, που πρέπει να υπάρξει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο και γι' αυτό, και καταλαβαίνετε τη δυσκολία, το καλοκαίρι εγώ θα υποβάλω την πρόταση βάσει του άρθρου 89 για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη με ρωτήσατε αν γνωρίζουν το πρόβλημα. Ήταν ένα άλλο ερώτημα. Σας μίλησα για αυτό το ελβετικό τυρί που αντιμετωπίζουμε. Και εδώ απαντάω και στο ερώτημα του κυρίου Ντεγιάνγκ. Πώς μπορεί να διώξει ένας ε, εθνικός ε, εισαγγελία αν δεν προβλέπεται τίποτα στην εθνική ένομη τάξη. Συχνά δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους εισαγγελείς για κακή πρόθεση ότι δεν κάνουν τίποτα για να υπερασπίσουν τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω της εθνικής νομοθεσίας τους. Δεν, προβλέπει, δεν, δεν προβλέπει καμία δράση για αυτού. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια κοινή βάση, ούτω ώστε οι εθνικοί εισαγγελείς να μπορούν να δρουν. Στη μελέτη αντικτύπου για την οδηγία κατά της απάτης που υπάρχει ήδη μπροστά μας, γιατί προφανώς χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να κάνουμε μια νομική πρόταση. Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι διαφορές στους ορισμούς καθιστούν αδύνατον μερικές φορές ή δύσκολο για τις εθνικές αρχές να διώκουν Ακριβώς για αυτά τα παραθυράκια και τις τρύπες σας μιλούσα προηγουμένως. Ο κύριος Νιούτον Ντάν πάει ένα βήμα παραπέρα και ονειρεύεται την Ευρώπη του μέλλοντος. Δεν είμαι σίγουρη ότι εσείς και εγώ θα κάνουμε ακόμα πολιτική όταν αυτή η νέα Ευρώπη γεννηθεί. Αλλά είμαι σίγουρη ότι και εγώ και εσείς θα ετοιμάσουμε το έδαφος ούτως ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτή η νέα Ευρώπη. Και θα ξέρετε σίγουρα ότι μόνο μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας ένας επίτροπος μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες του. Πριν όλα αποφασιζόταν με ομοφωνία και όλα ήταν στα χέρια των κρατών μελών. Επομένως η συνθήκη της Λισαβόνας μας έδωσε τρομερές δυνατότητες να προχωρήσουμε. Αλλά δεν μας έχει δώσει και την απόλυτη εξουσία πρέπει να προχωρήσουμε βαθμιδών. Αλλά σίγουρα τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας κάποια μέρα θα ζήσουν αυτή την πραγματικότητα ενός ευρωπαϊκού FBI. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Κύριε Ντεγιάνγκ, απάντησε ήδη σε κάποια από τα ερωτήματά σας. Τώρα, να απαντήσω στα υπόλοιπα. Για το λόγο που μόλις εξήγησα, επί του ερωτήματος του κυρίου Νιούτον Ντάν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ω προ το πόσο μακριά θέλουμε να πάμε και πάμε. Γιατί προφανώ αυτό είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Κυρία Ματιέ, έχετε δίκιο που λέτε ότι πολλά από τα κράτη-μέλη δεν έχουν καν διαβάσει τη συνθήκη ή δεν γνωρίζουν, ίσω υπεύθυνοι τη διάβασαν, αλλά δεν συνειδητοποιούν τι ε, επιπτώσεις της συνθήκης συνθήκη Λισαβόνα σε όλου αυτού του τομεί γιατί ακριβώς είναι τελείω νέα αυτά τα πράγματα. Αλλά έχουμε δυνατότητες, χάρη στη συνθήκη αυτή, και συζητάμε, ναι, πολύ τακτικά στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και δικαιοσύνη. Ειδικά στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνη, γιατί οι περισσότερε από τι προτάσει μου υποβάλλονται προς τους υπουργού δικαιοσύνη. Και σας λέω ότι ακόμα και όταν είμαι απόλυτα εντός των ορίων της συνθήκης, ακόμα και τότε υπάρχει έλλειψη κατανόησης. Πολύ μεγάλη από διαφορετικά κρατημέλη. Ακόμα και όταν είμαι απόλυτα εντός των όσων προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Επομένως, προχωράμε βήμα-βήμα. Και γι' αυτό ακριβώς χρειάζομαι τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τη χρειάζομαι πολύ. Γιατί εσείς ως ευρωβουλευτές δεν κοιτάτε τόσο πολύ την νομική παράδοση σε κάθε χώρα. Κοιτάτε το συμφέρον της Υπήρου μας και των 500 εκατομμυρίων πολιτών μας και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Τώρα, οι ελάχιστες κυρώσεις. Όχι μόνο για ένα έγκλημα, αυτό που προβλέπει η συνθήκη, αλλά για όλα τα εγκλήματα που ανέφερα. Αυτό θα το κάνουμε κάποια μέρα, αλλά όχι σήμερα. Δεν έχει φτάσει ακόμα αυτή η μέρα. Αμοιβαία αναγνώριση. Επόμενο σημείο. Από τη στιγμή που ανέλαβα αυτή τη δουλειά, έκανα ό,τι μπορούσα, ούτω ώστε να υπάρξει αμοιβαία κατά αναγνώριση. Θα θυμάστε όλους τους δικονομικούς κανόνες που είχαμε για άτομα που είναι υπόδικα. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη αμοιβαία εμπιστοσύνη. Μόνο όταν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση. Και δεν μπορείτε ε, μέσω διαταγμάτων να εξασφαλίσετε την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Γιατί σίγουρα θέλουμε να σεβαστούμε και την εξαρτησία της δικαιοσύνη. Και δεν μπορούμε μέσω διατάγματων να, να πούμε όλες οι Δικαιοδοσίε θα εμπιστεύονται τα όσα κάνει η γειτονική χώρα. α πούμε, κάθε ένωμη τάξη θα εμπιστεύεται τα όσα συμβαίνουν στην, συμβαίνουν ένωμη τάξη τη άλλη χώρα. Όχι, αυτό θα δημιουργηθεί, θα αναπτυχθεί λίγο-λίγο χάρη στα νομικά στοιχεία που έχουμε υποβάλει. Ποινικέ κυρώσει, διοικητικέ κυρώσει. Τα τη αυτά και λαμβάνοντα υπόψη και προτάσει τη δική σα έκθεση, κύριε Ντε Μια ομάδα επαϊόντων για τον ποινικό κώδικα για παράδειγμα, με στόχο να εξεταστούν όλα αυτά τα θέματα και να υποβληθούν σαφέστερες προτάσεις, να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε Είμαι ιδιαίτερα προσεκτική. Δεν είναι έτσι. Δεν αυτό σχεδιάζουμε κάποιες προτάσεις. Μελετώ τα πράγματα προτού υποβληθούν κάποιες προτάσεις. Μόνο όταν έχουν αντιμετωπιστεί τα θέματα της αντιμετώπισης ε, και της κατάστασης σε σχέση με τα κράτη-μέλη μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Έχω και νομίζω αυτό ήταν το ερώτημα από πλευρά συναδέλφου. Απάντησα σε σχέση το πότε και για την δημόσια συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση. Ναι, θα είναι πιο εύκολο να ε, αυξηθεί η συνειδητοποίηση των πολιτών και πολιτική η συνειδητοποίηση ε, και ίσως αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να υπάρξει η συνειδητοποίηση από πλευρά των πολιτών που θα πιέσει και θα προωθήσει τις εθνικές κυβερνήσεις στο να συμφωνήσουν και να αναλάβουν δράση. Και έτσι λοιπόν έτσι αντιμετωπίζω αυτή την πρότασή σας την οποία δέχομαι για την διοργάνωση μιας συνδιάσκεψης ενός, ε, ε, μιας διάσκεψης ε, και λαμβάνω υπόψη αυτή την πρότασή σας. Και εσείς κυρία Βάιλερ έχετε απόλυτο δίκιο επίσης. Η πυρωτική εντός εισαγωγικών διάσταση αυτών των συστημάτων. Η οικονομική διάσταση π.χ. Ε, από πλευρά ΗΠΑ υπάρχουν δυσκολίες να αντιμετωπιστεί το εμβαλωματικό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης οικοδόμημα και εδώ πρέπει να υπάρξει μια εντονότερη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά πρέπει να προχωρήσουμε με βάση τις ευρωπαϊκές συνθήκες εμείς οι Ευρωπαίοι και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τώρα θα ενσωματώσουμε, θα εντάξουμε την οικονομική, το οικονομικό έγκλημα σε αυτές τις δραστηριότητες ή όχι. Πιστεύω ότι απλά το γεγονός ότι η οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος έχει τεθεί στο τραπέζι από τον Μισελ Μπαρνιέ Επίτροπο στοχεύει προς την ορθή κατεύθυνση των εργασιών μας εδώ και το δείχνει αυτό για τις επαφές με τα κράτη-μέλη. Νομίζω έχω επεξηγήσει ε, σχετικά το, τις δυσκολίες που υπάρχουν καμιά φορά. Τώρα, τι κάνουμε σε σχέση με τα υφιστάμενα θεσμικά όργανα, με τους σήμερα εν λειτουργία θεσμούς και όργανα, OLAF, Europol, Eurojust, με όλα αυτά τα όργανα. Επεξήγησα ότι για τη δημιουργία του EPPO αυτό που θα κάνουμε είναι θα προτείνουμε, θα θέσουμε στο τραπέζι επίσης και τη μεταρρύθμιση την αναθεώρηση της Eurojust ώστε η εσωτερική δομή να είναι σαφέστερη και πιο αποτελεσματική από πλευράς Eurojust και να επιτρέπει επίσης και την αξιολόγηση από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων όλων αυτών, όλων αυτών των δράσεων. Αναφέρεται και στη συνθήκη ότι το μέσο αυτό, το EPPO, απορρέει αντλείται, προέρχεται από την Eurojust. Πρέπει λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία εκ παραλίλου να βαίνουν και να αναπτύσσονται, ώστε να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο και να προχωρήσουμε. Γνωρίζετε όμως ότι δεν έχει δυνατότητες ανακρίσεων ε, η Eurojust. Θα είναι διαφορετική σε σχέση με την EPPO όσον αφορά αυτή τη συνιστόσα. Όμως η Eurojust μπορεί να εξετάσει πάσης φύσεως εγκλήματα και παρατυπίες, όχι μόνο αυτά τα οποία βρίσκονται στη συνθήκη μας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ εξειδικευμένοι και πολύ εκλεπτισμένοι από πλευράς ε, συνεργασίας ε, που θα αναλυθεί και δραστηριοτήτων για την Όλαφ. Εξετάζουμε τις δυνατότητες διασύνδεσης Όλαφ και EPPO. Είναι όμως πολύ πρώιμη η χρονική στιγμή, πολύ νωρίς τώρα να πούμε και να δούμε πώς η Όλαφ θα ενταχθεί ή θα συνδέεται και πώς επίσης και η PPO θα εργάζεται και θα λειτουργεί σε σχέση με την Europol. Ένα πράγμα όμως είναι απόλυτα σαφές ήδη σήμερα. Η ΠΠΟ, η PPO θα εξετάζει τις ε, εγκληματικές ε, ανακριτικές δραστηριότητες ε, όπως και από τα ερωτήματα κιόλας απορρέει ότι έχουμε πάρα πολύ ευαίσθητα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν από πλευράς μας προτού υποβληθεί πρόταση στους αρμοδίους στο τραπέζι. Ο κύριος Γιακολίνο έκανε επίσης λόγο και για το ξέπλυμα ε, ε, χρημάτων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και σε σχέση με την πρόταση του ε, Επιτρόπου Μισελ Μπαρνιέ ανέφερα τα σχετικά και έχω ήδη και με άλλη μου παρέμβαση δώσει ε, κάποια στοιχεία. Η κυρία Γιώτοβα έκανε μια παρέμβαση για την έκθεση της ε, μονάδας κατά της διαφθοράς. Είναι στα χέρια της συναδέλφου μου επιτρόπου Σεσίλια Μάνστρομ το θέμα αυτό και σίγουρα εκείνη θα προσέθει και θα εκθέσει στους ευρωβουλευτές εδώ στην Ευρωβουλή τα σχετικά. Γνωρίζετε ότι το, θέμα επίσης της διαφθοράς εγγράφεται, βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της έκθεσης CVN και είναι ο Γενικός Γραμματέας που θα δίνει συνέχεια σε αυτά τα θέματα και για τη Ρουμανία και για τη Βουλγαρία καθώς η διαφθορά είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία πάνω-πάνω στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα συνεχίσουμε με το δεύτερο πάνελ, την αναδιάρθρωση της Europol και της Eurojust για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και του χρηματοοικονομικού διασυνοριακού εγκλήματος. Προοπτικές για μια ευρωπαϊκή FBI. Ε, θα μιλήσουμε τον κύριο Γιώργ ο οποίος είναι υπεύθυνο του de l'Europe, που θα μας μιλήσει για το ρόλο της Europol και της Eurojust και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και θα ε, συνομιλήσουμε τον κύριο Έρικ Μπάρνετ εντεταλμένο του από το Υπουργείο Εξωτερικών, Εσωτερικών με συγχωρείτε, τον ΙΠΑ. Ε, Όσον αφορά την ε, διαδικασία θα έχουμε μία παρουσίαση ε, από τον κύριο Μονάρ και μετά από τον κύριο Μπάρνετ και μετά ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές. Με προτεραιότητα των, ε, τους εισηγητές των πολιτικών ομάδων καθώς και τους υπεύθυνους από τις Επιτροπές ΛΥΜΠΕ και ΚΡΙΜ. Ε, κύριε Μονάρα, έχετε το λόγο. Uh, uh, um, Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και μπορώ να συγχαρώ οπωσδήποτε την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και κρίμα για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας διότι η πρόκληση αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος δεν υπάρχει νομίζω επαρκώς πάντα στα μέσα διότι συνήθως εστιάζονται στα θέματα τρομοκρατίας όμως πάρα πολλές ζωές, περισσότερες ζωές χάνονται ετήσια λόγω των διαστάσεων του οργανωμένου εγκλήματος ε, σαν αποτέλεσμα. Τώρα, σε σχέση με το θέμα, συγκεκριμένα ο ρόλος Eurojust Europol, Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι πιστεύω ότι αυτά τα θεσμικά όργανα, αυτές οι υπηρεσίες ήδη συνεισφέρουν με μείζωνα τρόπο για την καταπολέμηση, στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και αυτό όχι μόνο λόγω της υποστήριξης που παρέχουν στις εθνικές αρχές ε, υπό τους όρους ε, διαδικτύωσης, υποστήριξης ε, σε δίκτυα ή και τεχνικά, αλλά επίσης επειδή διαδραματίζουν ένα πολύ ενεργό ρόλο στο ίδιο το πεδίο στη δράση τους και πρέπει κανείς να ταυτοποιήσει δύο συνιστώσεις, δύο παραμέτρους. Η, πρώτη είναι ότι αυτές οι δύο οργανώσεις, αυτές, αυτά τα δύο όργανα διαδραματίζουν ένα συντονιστικό ρόλο ήδη σήμερα. Μπορούν να δώσουν προσανατολισμούς προς τις αρχές, ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς που πριν από τη δημιουργία τους δεν υπήρχαν. Και από πλευράς Europol ιδιαίτερα βλέπουμε ότι δίνεται μια σημαντικότατη συνεισφορά για την αντιμετώπιση των κοινών στην προσέγγιση τους κινδύνων που πρέπει να αντιμετωπιστούν διότι χωρίς αυτή την κοινή προσέγγιση δεν μπορούν να τεθούν προτεραιότητες στην ημερήσια διάταξη για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και υπάρχει ιδιαίτερη πρόκληση της ε, εφαρμογή του νόμου και τη συμμόρφωσης με αυτές τις πτυχές. Δεν υπάρχει κανένα άλλο θεσμικό όργανο που από πλευρά του δομής του να μπορεί να παράσει τέτοιου είδους ε, ε, δραστηριότητες και δυνατότητες και υπό τους, ήρους, υπό τους όρους της ανάπτυξης της Eurojust και της Europol περαιτέρω μεταξέλιξης πρέπει να συνειδητοποιήσει κανείς και τις τους περιορισμούς που η συνταγματική δομή προκαλεί και δημιουργεί για αυτές τις δύο υπηρεσίες διότι η εσωτερική ασφάλεια άρθρο 4 η εδάφια 2 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης όπως αναφέρεται είναι κύριο έργο που πρέπει να σέβεται από πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα κράτη-μέλη και θέτει σαφείς περιορισμούς για τις δράσεις της Europol η συνθήκη και βλέπουμε εδώ ότι τα μέτρα κύρωσης ε, εξακολουθούν να είναι κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω και κάτι, καθώς όλα αυτά εντάσσονται υπό τον τίτλο των προοπτικών για την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας ως το FBI, ακόμα και αν δεν υπήρχαν αυτοί οι περιορισμοί από πλευρά σας συνθήκης, θα είχαμε κάποιες πολύ σημαντικές επιφυλάξεις που θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη. Επιφύλαξη πρώτον συνταγματικού χαρακτήρα, συνταγματικής φύσεως. Αν συγκρίνουμε την ευρωπαϊκή δομή με την δομή των ΗΠΑ υπάρχει σαφώς ε, το FBI που εργάζεται και λειτουργεί υπό τις ε, αρμοδιότητες και εντολές του Προέδρου πλήρως ε, δημοκρατικά σε ε, μια τέτοια πολιτιακή δομή. Εμείς όμως δεν έχουμε μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση που να μπορούσε να δίνει μια τέτοια, ένα τέτοιο πλαίσιο ε, ένταξης και κατοχήρωσης αυτών των αρμοδιοτήτων αυτής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας. Και θα χρειαζόταν μια νέα συνθήκη για την κατανομή των εξουσιών και των κυριαρχικών δικαιωμάτων για την καταπολέμηση του εγκλήματος που δεν προβλέπεται και δεν παρέχεται από τη συνθήκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Ένα τρίτο ως επιφύλαξη είναι ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πλούτο πολυμορφίας όσον αφορά διαφορετικούς πολιτισμούς ε, πολιτιακούς, ε, δικαστικούς, επιβολής δικαίου, ποινικού και αν δημιουργούσαμε μια υπερεξουσία αυτό θα αντιμετώπιζε, αυτή η προσπάθεια θα αντιμετώπιζε αμέσως πολλές αντιστάσεις ε, από πάμπολες πλευρές. Λοιπόν, δεν λέω ότι είναι ανέφικτο ή αδύνατο να υπάρξει μια τέτοια δυνατότητα μια τέτοια υπηρεσία, αλλά θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Όχι μόνο χρόνο για την αλλαγή συνθήκη, αλλά και για την αλλαγή τη νοοτροπία. Και η αλλαγή νοοτροπία τι πιο πολλέ φορέ χρειάζεται το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Να πω και δύο λόγια τώρα, παρότι γνωρίζω ότι αυτό είναι θέμα για την επόμενη διάσκεψη, τον επόμενο γύρο, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό έχει τη σπουδαιότητά του ω θέμα και για τη δική μα ε, συνεδρίαση και το δικό μα γύρο. Διότι αν δημιουργηθεί μια τέτοια εισαγγελία με τέτοιου είδους ε, ε, εξουσίες ε, θα μπορούσε να υπάρξει μια ας το πω έτσι μια δυνατότητα που θα έπρεπε να μπορέσουμε να συγκεράσουμε διάφορες ας το πω έτσι αντικρώμενες απόψεις γεφυροποιώντας τα πράγματα ένας ε, δεσμός μεταξύ της ε, δημιουργίας του EPPO και της ε, δημιουργίας της δυνατότητας των εξεταστικών ανακριτικών εξουσιών. Αυτό δεν επιλύει αυτόματα όμως τα θέματα τα οποία σας προανέφερα προηγούμενα υπό τους όρους της γενικότερης συνταγματικής δομής ως διάρθρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα προβλήματα που δημιουργούνται. Υπάρχει όμως εδώ ένα συνδετικός κρίκος, ένα κομβικό σημείο. Όμως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένα μείζον εγχείρημα ίσως το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο εγχείρημα σε αυτή τη χρονική συγκυρία στον χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας, διότι για πρώτη φορά υπάρχει αυτή η προοπτική του συνδυασμού δικαστικών αρμοδιοτήτων και αστυνομικών διοκτικών δικαιωμάτων και δυνατοτήτων. Και βλέπω να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος κίνδυνος εδώ. Αν επενδυθεί υπερβολικό κεφάλαιο πολιτικά ε, στο εγχείρημα του EPPO και έχουμε άλλες δομές που μπορεί ίσως να παραμεληθούν ή άλλες πτυχές που θα μπορούσαν να παραγνωριστούν και να αμεληθούν, να μην ξεχνάμε ότι από πλευράς αυτού του γραφείου, αν θεσπιζόταν, θα είχε περιορισμένο εύρος εντολής. Θα ήταν η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα κλάσμα δηλαδή μόνο, ένα μικρό τμήμα όλων των δραστηριοτήτων δίωξη εγκλήματο που θα μπορούσαν να καλύπτονται υπό αυτή την εντολή. Και βλέπουμε εδώ και το τι θα ε, ε, πρέπει να γίνει σε σχέση με τη συμμετοχή άλλων όπως π.χ. Βρετανών και ε, άλλων σε αυτή την πρωτοβουλία. Υπάρχουν ίσω εδώ λιγότερο ενθουσιώδεις πρόπτικες. Όμως, δίνοντα συνέχεια σε αυτή την εναλλακτική δυνατότητα θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και άλλε πτυχέ πτυχές, άλλες δυνατότητες όπως την ενίσχυση της Eurojust και την ενδυνάμωση και της Europol. Πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν. Λοιπόν, στην περίπτωση της Eurojust πρώτον, νομίζω η συνθήκη διανοίγει την δυνατότητα να ε, έχουμε την Eurojust με εξουσίες που θα αναλάβει όσον αφορά την έναρξη ανακριτικών δραστηριοτήτων και διοκτικού έργου και με δεσμευτικές αρμοδιότητες όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων αντικρουωμένων συμφερόντων και τριβών μεταξύ δικαστικών αρχών μεταξύ των κρατών μελών μας. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τύχει της προσοχής μας και συνεργασία και με τις δικαστικές αρχές. Διανοίγει η συνθήκη δυνατότητες που θα έπρεπε πολύ σοβαρά να εξετάσουμε ιδιαίτερα με τη στην δημιουργία του ΕΠΠΟ που γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο και θα έχει περιορισμένο ε, εύρος εμβέλειας εντολής. Επίσης εδώ υπάρχει ένα δυναμικό για την καλύτερη χρήση πραγματογνωμοσύνης ε, της Eurojust ε, για την καταπολέμηση μιζώνων μορφών οργανωμένου εγκλήματος. Αυτή τη στιγμή η επικέντρωση είναι η χρήση των αναλυτικών εργαλείων και μέσων της Europol. Eurojust όμως από την άλλη πλευρά βρίσκεται και εκείνη στον, στην πρώτη γραμμή με τόπου στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Και αυτή η πτυχή λοιπόν θα πρέπει να τύχει καλύτερη εκμετάλλευση, καλύτερη χρήση στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η συνέργεια μεταξύ Eurojust και Europol θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί διασφαλίζοντας ότι Eurojust θα μπορεί να συμμετάσχει σε όλες τις ε, δραστηριότητες Europol. Αυτή η συνεργασία και συνέργεια μεταξύ των δύο αυτών οργάνων Europol και Eurojust πρέπει να μεγιστοποιηθεί και να βελτιστοποιηθεί. Για την Europol υπάρχει σημαντικό δυναμικό για την ανάπτυξη του ε, δυναμικού αξιολόγησης ε, της Europol, διότι βρίσκεται σε στρατηγικά πάρα πολύ αξιόλογο κομβικό σημείο να μπορούμε να δούμε πώς η δράση των κρατών μελών ανταποκρίθηκε στον εντοπισμό και ταυτοποίηση των μεγαλύτερων προκλήσεων του οργανωμένου, από πλευρά οργανωμένου εγκλήματος. Ένα πίνακα επιδόσεων δηλαδή. Ένα θέμα είναι ο εντοπισμό και ταυτοποίηση των μιζώνων μορφών ε, οργανωμένου εγκλήματος, αλλά αυτό αποσυνδέεται από το με πόσο καλό τρόπο αντιδρούν, αντιδρούν τα κράτη-μέλη και αναλαμβάνουν δράσεις για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, κατονομάζοντας σαφώς εκείνα τα κράτη και εκείνες τις αρχές που δεν λειτουργούν όπως πρέπει και δεν έχουν καλές επιδόσεις. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υποβάλλονται αξιολογήσεις με παραρτήματα που θα μας δίνουν τη δυνατότητα να δούμε ποια κρατημέλη αποτυγχάνουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέσα. Γιατί να μην αυξήσουμε την πίεση λοιπόν στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος κάνοντας, αναλαμβάνοντας τέτοιου είδους δράσεις όπως αυτή σε σχέση με τις επιδόσεις χρειαζόμαστε και καλή, ε, καλό επίπεδο κατανόησης όσον αφορά το κόστος ε, σε ανθρώπινο δυναμικό. Ε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο λιτότητας και περικοπών. Σε μια τέτοια περίοδο δεν μπορεί όλοι οι στόχοι να ακολουθούνται ταυτόχρονα εξίσου ισοπεδωτικά. Πρέπει να έχουμε προτεραιότητες για το τι πρέπει να γίνει πρώτα και τι πρέπει να γίνει έπειτα. Πρώτα τα ουσιώδη σε άλλη φάση, σε ακόλουθη φάση τα λιγότερο ουσιώδη. Πρέπει να εστιαζόμαστε στις κυριότερες προκλήσεις και έτσι να δρούμε, βλέποντας τι απορρέει ως κύριο συμπέρασμα στις δράσεις μας σε όλους τους ε, τομείς, σε όλα τα πεδία και ποιο είναι το κόστος που συνεπάγονται αυτές οι δράσεις, ενδυναμώνοντας επίσης και τον ρόλο της Europol. Όσον αφορά την ε, έναρξη, το σχεδιασμό, την υλοποίηση κοινών αστυνομικών δράσεων. Αυτή τη στιγμή μπορεί να υποβάλει προτάσεις η Europol, να αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλλά δεν έχει ιδιαίτερα δραστήριο ρόλο για την υλοποίηση και εκτέλεση όλων αυτών των κοινών αστυνομικών δράσεων. Και νομίζω έχουμε εδώ ένα πεδίο στο οποίο τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Με τη Frontex για παράδειγμα και με την υπηρεσία ΣΥΛΟΥ, θα υπάρχουν ομάδε με ε, κρατικού υπαλλήλου από τα κράτη-μέλη που θα μπορούν με το βέλτιστο τρόπο να εκμεταλλευόμαστε. Pools δηλαδή κοινέ ομάδες ε, με διαφορετική σύνθεση από τα κράτη-μέλη και τα όργανα αυτά για να έχουμε τη βέλτιστη επίδοση. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, η τελευταία μου παρατήρηση επ' αυτών είναι μια παρατήρηση που συνδέεται με την χρηματοδότηση, τα οικονομικά, τα κονδύλια. Οποιαδήποτε περαιτέρω ενδυνάμωση της Eurojust και της Europol έχει αυτή τη συνέπεια. Αυτά που βλέπουμε τώρα σε αυτή τη φάση είναι ουσιαστικά συστηματικές πολιτικές περικοπών όσον αφορά τα κονδύλια για αυτές τις υπηρεσίες. 82 εκατομμύρια έχει η Europol σε ε, κονδύλια που προβλεπόντουσαν που περικόπησαν σε 75 εκατομμύρια τώρα για το, το κυβερνο, κυβερνοέγκλημα που εντάσσεται και αυτό στις δραστηριότητες της Europol θα έπρεπε να είχαμε περισσότερα κονδύλια και όχι λιγότερα. Είναι μια σχιζοφρενική, παρανοϊκή κατάσταση αυτή που σημειώνεται σε σχέση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Αφενός δίνουν όλο και περισσότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες σε αυτές τις υπηρεσίες και αυτό ε, ισχύει και για τη Eurojust. Ταυτόχρονα όμως από την άλλη πλευρά περικόπτουν κονδύλια. Υπάρχει μια πολύ καλή ε, τοποθέτηση ως απόφθεγμα σε περιόδους ε, κρίσεων θα πρέπει κανείς με λιγότερα χρήματα να κάνει περισσότερα. Ωραία ακούγονται όλα αυτά, αλλά υπάρχουν περιορισμοί αγαπητοί ευρωβουλευτές σε τέτοιου είδους εγχειρήματα. Επίσης ε, είναι σωστό αυτό το οποίο λέγεται ότι παίρνεις αυτό που πληρώνεις, πληρώνεις λιγότερα, θα έχεις ε, μικρότερο αποτέλεσμα και λιγότερα αποτελέσματα. Να ληφθεί και αυτό υπόψη. Κάθε ευρώ που επενδύεται στον προπολογισμό αυτών των υπηρεσιών έχει αποτέλεσμα πολλαπλασιαστικό για τα ωφέλη που απορρέουν για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Αυτές οι υπηρεσίες είναι πραγματικά μέσα και εργαλεία έκφρασης ευρωπαϊκά της αλληλεγγύης. Διότι δίνουν υποστήριξη, αρρωγή στα κράτη-μέλη που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια για να απαντήσουν και να αντιδράσουν στην πρόκληση του οργανωμένου εγκλήματος στο οργανωμένο έγκλημα. Ό,τι μπορείτε εσείς λοιπόν ευρωβουλευτές ε, να πράξετε για να αντιμετωπιστεί η ορθή, η δίκαια αντιμετώπιση αυτών των οργάνων, αυτών των θεσμών θα είναι ευπρόσδεκτο για να είμαστε στο ύψο των περιστάσεων. Σα ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Μονάρ, είναι πολύ δύσκολο το έργο αυτό. Είμαστε όλοι θύματα τη ε, λιτότητα και όμω έχουμε τόσα πολλά μέτωπα ανοιχτά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπάρνετ. που είναι επιτετραμένος ε, του Αμερικανικού Υπουργείου Ιστορικής Ασφάλειας και των, του Τμήματος Ερευνών και ανήκει στην, είναι αποσπασμένος εδώ στην Αμερικανική Διπλωματική Ομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Θέλουμε να σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δείτε να κάνουμε μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων για την, ε, τον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Είμαι επιτετραμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση α, από την ε, Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνίων. Ε, έχει το ακρονίμιο ICE. Πριν από αυτό, επί 15 χρόνια ήμουν εισαγγελέα και τα μισά αυτά χρόνια ήμουν σε επίπεδο πολιτείας ε, τα υπόλοιπα χρόνια ήμουν ομοσπονδιακό ε, εισαγγελέα στο Υπουργείο Δικαιοσύνη των ΗΠΑ. Το ISIS ε, είναι τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που δημιουργήθηκε μετά την τρομοκρατική επίθεση τη της 10 Σεπτεμβρίου. Έχει ερευνητικές αρμοδιότητες μαζί με τις μεταναστευτικέ υπηρεσίε και τι τελωνιακέ αρχέ. που ήταν η παλαιότερη, η παλαιότερη υπηρεσία στι ΗΠΑ, το 1979 δημιουργήθηκε. Εμείς έχουμε 4,5 εκατομμύρια ευρώ ε, προϋπολογισμό και ε, επίσης ε, έχουμε ειδικούς πράκτορες 7.000 για τις έρευνες αυτές. Έχουμε 200 γραφεία στις Ηνωμένε Πολιτείες και γραφεία σε 49 χώρες, καμιά εβδομηνταριά ασχολούμαστε με την διερεύνηση του ε, διεθνούς εγκλήματος. Επίσης, υπάρχουν πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες ε, διοκτικών αρχών, ε, το FBI, DA, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλες ε, υπηρεσίες που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Εγώ δεν εκπροσωπώ αυτές τις υπηρεσίες, αλλά είναι βασική στρατηγική εταίρη. Σε ό,τι αφορά το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, το, η υπηρεσία μου είναι μια ε, διασυνοριακή ερευνητική υπηρεσία. Ε, προσπαθούμε να δούμε ε, πώς χρηματοδοτείται το παράνομο εμπόριο ε, προς και από τις ΗΠΑ. Συχνά υπάρχει υπόθεση ότι οι διοκτικές αρχές της ΗΠΑ ε, ερευνούν τα περισσότερα εγκλήματα. Όμω, ένα μικρό ποσοστό των εγκλημάτων στι ΗΠΑ διερευνάται από τι ομοσπονδιακέ ε, διοκτικέ αρχέ. Οι περισσότερε ε, αρχέ που ερευνούν τέτοια εγκλήματα είναι πολιτιακέ αρχέ. Όμω, η HSI, η δική μου υπηρεσία, έχει μια ε, εθνική δια... αρμοδιότητα και υπερεθνική και μπορεί να δώσει και πόρους, τι έρευνες και πραγματογνωμοσύνη ε, να σας δώσω παραδείγματος χάρη. Ε, οι ειδικοί πράκτορες του HSI ε, μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 ε, συνέλαβαν 29.000 άτομα για ομοσπονδιακά εγκλήματα. Ε, για διεθνικό έγκλημα, ε, λαθρεμπόριο στι ΗΠΑ, ε, λαθρεμπόρια, παραδείγματο χάρη για την παραχάραξη αγαθών, μαϊμούδε κτλ. Για εμπόριο ανθρώπων, ε, σεξ, ε, σεξουαλική εκμετάλλευση, και γιατί το λαθρεμπόριο μέσω των συνόρων σημαίνει ε, ότι μπαίνουν αγαθά και βγαίνουν αγαθά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε εδώ και για όπλα, για τη στρατηγική τεχνολογία. Ε, πολλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να κατασκευαστούν όπλα μαζικής καταστροφής από αυτά τα υλικά. Επίσης, άλλες ε, διοκτικές αρχές έχουν αντίστοιχες στατιστικές συλλήψεων, αλλά καμία αρχή Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορεί να πετύχει την αποστολή της χωρίς καλές Σχέσει με τις άλλες υπηρεσίες. Στι ΗΠΑ αυτό το καταφέρνουμε μέσω τη δημιουργία ομάδων κρούσεων, task force, που επιτρέπουν στι ομοσπονδιακέ αρχέ να ομαδοποιήσουν φόρου ε, την πραγματογνωμοσύνη ε, σε ομοσπονδιακό επίπεδο και να χρησιμοποιήσουμε και ό,τι πόρου υπάρχουν σε πολιτιακό επίπεδο. Και ο στόχο είναι να καταπολεμήσουμε μια συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα με όλο το πλωστάσιο των πόρου έχουν τη δικαιοδοσία, τα, τις ικανότητες που έχουν οι πολλαπλές υπηρεσίες. Το HSI συμμετέχει σε πολλές task force υπό την αιγίδα άλλων υπηρεσιών. Παραδείγματο χάρη στην Task Force ε, για, τα, για το λαθρεμπόριο ε, ναρκωτικών, ε, για την εκμετάλλευση των παιδιών, α πούμε, μια άλλη κτλ. Επίσης η HSI ηγείται διαφόρων τέτοιων ομάδων κρούσεων ε, το κέντρο, ας πούμε, κυβερνο, για το κυβερνοχώρο λοιπά. Έχουμε μία task force όπου συμμετέχουν 17 ε, αμερικανικές υπηρεσίες, ε, η Interpol, η Europol λοιπά. Στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, προσπαθούμε να δούμε οι διεφθαρμένοι ε, υπάλληλοι πώς ε, πώς ε, βοηθούν στην, στο ξέπλυμα του χρήματος. Άλλες task force ε, τις διαχειρίζεται η, η HSI στη Νέα Υόρκη και εκεί έχουμε 55 διοκτικέ αρχές που συμμετέχουν. Αυτή η Task Force ε, συνεργάζεται με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ε, χρησιμοποιεί ε, παρακολουθήσεις, παρακολουθήσει, email, καθώς και διάφορες πληροφορίε. και αυτό έδειξε ότι η HSBC δεν μπόρεσε να εφαρμόσει ελέγχους κάτι του ξεπλήματο του χρήματο, η τράπεζα αυτά, και γι' αυτό ήρθε σε ε, χρειάστηκε να την τιμωρήσουμε ε, με ένα ποσό, έδωσε λέει στις ένα ποσό 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. η διασυνοριακή, το συνεδριακό λαθρεμπόριο χρηματοδοτεί τις εγκληματικές οργανώσεις. Υπάρχουν μια πλειάδα εγκληματικών δραστηριοτήτων και με αυτόν τον τρόπο προχωρούν στις δραστηριότητές τους οι εγκληματίες αυτοί. Επειδή ακριβώς ε, υπάρχει αυτή η αρχή ότι το χρήμα κινεί τα πάντα, δημιουργήθηκε αυτή η ειδική task force που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, ε, για να ηχνηλατήσει, ανιχνεύσει ε, την διακίνηση του χρήματος. Αυτός ο φορέας προβαίνει και σε κατασχέσεις ε, σε περίπτωση ε, λαθρέας ε, μεταφοράς χρημάτων και ούτω καθεξής. Η διεθνής εφαρμογή του δικαίου δεν μπορεί να εφαρμοστεί κατά τον ίδιο τρόπο όπως ισχύει με τις δικές μας task forces. Θα πρέπει να υπάρχουν επιτόπου μηχανισμοί που να συντονίζουν την πολυμερή συνεργασία ε, υπήρξε ε, μία ε, συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου καταπολέμησης του εγκλήματος στο κυβερνοχώρο από πλευράς Ευρώπης και από πλευράς ΗΠΑ. Αυτά τα κέντρα θα ανταλλάξουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με θέματα απάτης, εκμετάλλευση των παιδιών και ε, με τις διοκτικές αρχές και από τις δύο πλευρές ως προς την εκμετάλλευση των ε, ανηλίκων. Πρόκειται για μια εγκληματική δραστηριότητα που έχει διεθνικό χαρακτήρα γιατί υπάρχει και δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου έτσι ώστε να περνάμε τα ε, σύνορα ταχύστα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ε, σε αυτούς τους εγκληματίες να συνεχίσουν την ε, εγκληματική τους δραστηριότητα. Γι' αυτό αυτός ο φορέας, ο EC3 και ο C3, δηλαδή η συνεργασία τα γραφεία από πλευράς ΙΠΑ και Ευρώπης, προβάλλουν αυτή τη συνεχή συνεργασία με το δικό μας φορέα οι αρχές της ε, Δανίας ε, μπόρεσαν να ανοιχνεύσουν ένα room όπου φαινόταν ότι ένα ανήλικο αγόρι ήθελε να ε, βιάσει ένα ενδεκάχρονο κορίτσι και ε, σε αυτή την περίπτωση υπήρχε και μία ε, εικονογράφηση, δηλαδή ένα ηλιοτρόπιο το οποίο είναι χαρακτηριστικό στους δρόμους του Κάνσας. Και έτσι καταφέραμε να σώσουμε το παιδί λίγα λεπτά πριν βιαστεί, γιατί ανοιχνεύσαμε αυτό το χωριό. Έτσι οι διοκτικές αρχές της ε, Δανίας κατάφεραν να ιχνηλατήσουν αυτό το έγκλημα λίγα λεπτά πριν ε, διαπραχθεί. Γι' αυτό η δίωξη θα πρέπει να ε, βασίζεται σε όλα τα στοιχεία σε σχέση με τον βιασμό ή την απόπειρα βιασμού ανηλίκων παιδιών. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε ροή πληροφοριών από τις ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε καταδίκη ενός ατόμου για πορνογραφία με βάση βίντεο που έδειχναν έναν ενήλικα ο οποίος ε, βίαζε και κακομεταχειριζόταν ένα 18 μωρό. Είδαμε ότι αυτή η εγκληματική δραστηριότητα ε, έλαβε χώρα στην Ολλανδία. Σε αυτή την περίπτωση ε, υπήρξε και ομολογία αρκετών τέτοιων εγκλημάτων σε έναν βρεφονιπιακό σταθμό. Έτσι μπορέσαμε να σώσουμε πολλά παιδιά σε 60 σημεία ανά τον κόσμο. Αυτή, αυτή η δίωξη των, ε, των βιασμών ή της απόπειρας βιασμού ανηλίκων έγινε εξαιτίας της συνεργασίας μεταξύ ΙΠΑ και Ευρώπης. Οι διοκτικές αρχές των ΙΠΑ και ο δικός μας πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε ότι θα πρέπει να μπορούμε άμεσα να συνεργαζόμαστε και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για καταπολέμηση του εγκλήματος τη στιγμή που δεν αναγνωρίζουμε το, το, το ζωτική σημασία ρόλο της ανταλλαγής πληροφοριών. Θα ήθελα εντάχει να σας πω για μια προσωπική ιστορία που δείχνει τις προκλήσεις στην δίωξη του διεθνικού εγκλήματος. Η μητέρα μου μετανάστευσε το 1956 από την Ουγγαρία στη ΣΥΠΑ και πρόσφατα μου είπε μία ιστορία όπου, εκεί όπου μεγάλωσε η γιαγιά μου. Ε, πρόκειτο για τον θείο μου το Γιώσκα, ο οποίος ε, ε, έζησε 100 χρόνια και μπόρεσε να μας μιλήσει για τη ε, ζωή του. Είπε λοιπόν ότι γεννήθηκε στην Αυστρία αλλά πήγε στο σχολείο στην Τσεχοσλοβακία ε, μετά παντρεύτηκε στην Ουγγαρία και εργάστηκε στη Σοβιετική Ένωση, μετά δε αποσύρθηκε στην Ουκρανία. Κάποιος είπε, μαθία Γιώσκα, δεν ξέραμε ότι είχες ταξιδέψει τόσο. Και ο θείος Γιώσκα απάντησε, εγώ ποτέ δεν έφυγα από αυτό το χωριό. Και αυτό δείχνει τις προκλήσεις, τις δικές μας προκλήσεις. Δηλαδή τα σύνορα αλλάζουν, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις χώρες είναι ίδιοι και ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ζουν θα πρέπει να μπορούν να ζουν χωρίς έγκλημα, χωρίς χρηματικό έγκλημα, χωρίς διαφθορά και χωρίς εγκληματικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις που δεν σέβονται τα σύνορα. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις κατακερματισμένες εθνικές κυριαρχίες έτσι ώστε να μπορέσουμε συλλογικά να προστατεύσουμε τους πάντες από την εγκληματική δραστηριότητα. Θα ήθελα να προσπαθήσω να σας απαντήσω κατά το δυνατόν και θα δεχτώ με μεγάλη χαρά τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε κύριε Μπάρνετ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν έχετε ερωτήσεις... Mr. Dunn. Well, well, first of all, to, to... Κύριε Ντάν, κύριε Μόναρ, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Φυσικά θα πρέπει να περάσουμε από διάφορες φάσεις, από διάφορα βήματα. Ε, τα περιγράψατε και ο σκοπός είναι η μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Στις, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο δεν συνεργάζεται καθόλου, είναι φρικόδες αυτό, είναι το πρόβλημα της χώρας μου. Βρίσκουμε επιχειρήματα και λέμε ότι α, οφείλονται, οφείλονται αυτή η αποστασιοποίησή μας ε, στις μνήμες, στις αναμνήσεις που έχουμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάπως πρέπει να ξεκολλήσουμε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μέλλον όλοι, να βρούμε τη θέληση για το μέλλον. Ε, διερωτώ με αν το κείμενό σα θα τα μοιραστεί. Γιατί αυτά που είπατε για το Frontex και για το άσυλο δεν τα ήξερα. Θα μπορούσατε να μα δώσετε περισσότερε πληροφορίε. Δεν είναι ερώτηση αυτή, έτσι, ένα αίτημα είναι. Για περισσότερε πληροφορίε. Κύριε Μπάρνετ, πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία του θείου σα. Η γυναίκα μου το 1956 μετανάστευσε από την Ουγγαρία. Στον Βασίλειο προφανώ. Καταλαβαίνω και ταυτίζομαι με, τα όσα είπατε. Ε, προσφερθήκατε να μας βοηθήσετε και στο ταξίδι που θα κάνει η αντιπροσωπεία μας στη Ουάσιγκτον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, πήρα σημειώσεις από την παρουσίασή σας. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε υπόθεμα χαρτιού, α πούμε, η παρουσίαση σας. Καταλαβαίνω ήταν άτυπη και η ερώτησή μου είναι άτυπη. Πάντως πρέπει, μπορούμε να μάθουμε πολλά από εσά. σα ευχαριστώ που θα μα βοηθήσετε στο ταξίδι που θα κάνουμε, ούπου. Σα ευχαριστώ ακόμα μία φορά. Thank you, Mrs. Κυρία Βάιλερ. ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich sagen. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Οι δύο παρουσιάσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Εμείς έχουμε κάποιες επικρίσεις, κάποιο σκεπτικισμό. Μερικές φορές είναι απογοητευτικό όταν βλέπουμε πόσες φιλοδοξίες έχουμε και πόσες λίγες πιθανότητες να τις υλοποιήσουμε. Κύριε Μπάρνετ, είπατε ότι πρέπει να κινηθούμε προς μια άλλη κατεύθυνση. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν, όλοι τις ξέρουμε. Ε, το θέμα δεν είναι μόνο το να δώσουμε χρήματα. Το θέμα είναι να ξεπεράσουμε και τις διαφορετικές νοοτροπίες. Εμείς έχουμε 16 lender στη χώρα μου. Και κάθε land έχει τη δική του ένωμη τάξη ουσιαστικά στη Γερμανία. Και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ακόμα και μετα... η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων lender είναι προβληματική. Θα θυμάστε το σκάνδαλο, θα έχετε ακούσει για το σκάνδαλο της έρευνας για το NSU. Και ακούσαμε ότι υπήρχαν πληροφορίες, υπήρχαν δεδομένα, υπήρχαν στοιχεία τα οποία τα κράτησαν και δεν τα ε, κοινοποίησαν σε αυτά, στα πλαίσια αυτής της έρευνας. Ήταν μια τεράστια έρευνα, ε, υπήρξαν πάρα πολλές δυσκολίες και βλέπω ότι τέτοιες δυσκολίες έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες. Έχω πάει στην ε, Ιταλία, στο Παλέρμο και στη Ρώμη και εκεί είδαμε ότι οι Ιταλοί έχουν καλά εργαλεία για την εφαρμογή του νόμου και για τις ε, έρευνες. Ε, μας λένε λοιπόν, εσείς γιατί στην ε, Γερμανία είστε τόσο απρόθυμοι να ακολουθήσετε κι εσείς αυτό το δρόμο. Γιατί ανησυχείτε τόσο πολύ. Ε, για θέματα ας πούμε υποκλοπών και τέτοια, παρακολουθήσεων και αυτά στην Ιταλία, επειδή ας αναγκάστηκαν να ερευνήσουν ε, τα εγκλήματα της μαφίας, ε, πολύ γρήγορα χρησιμοποίησαν τέτοια μέσα, τα οποία έδωσαν καρπούς. Ε, η Europol, η Eurojust και η Olaf είναι ακόμα σε εμβριακή φάση. Εμείς στη Γερμανία ακούμε θετικά πράγματα για αυτές τις υπηρεσίες και για τα όσα έχουν επιτύχει. όσοι συνεργάστηκαν με τις υπηρεσίες αυτές μιλάνε με τα καλύτερα λόγια. Αλλά αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα, δεν το αρνούμε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλοι έχουμε τα συμφέροντά μας να συνεργαστούμε. Όλοι και εμείς. Όλοι μας πρέπει να συνεργαστούμε. Γιατί το οργανωμένο έγκλημα ανθεί σε μια εποχή οικονομικής κρίσης το οικονομικό έγκλημα αναπτύσσεται με τρόπους που 10-15 χρόνια πριν δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Και χάρη στο ίντερνετ και χάρη σε όλες τις υπόλοιπες τεχνολογικές εξελίξεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, ζούμε σε μια τελείως διαφορετική εποχή από ότι 20 χρόνια πριν. Γι' αυτό λοιπόν όλοι έχουμε συμφέρον να καταπολεμήσουμε αυτό το έγκλημα. Γιατί πραγματικά είναι απώλεια από το δημόσιο κορβανάο τα χρήματα αυτά που μπαίνουν στις τσέπες των εγκληματιών. Και αν δείτε, το λαθρεμπόριο τσιγάρων, ακόμα και στι ΗΠΑ μιλάμε για ποσά που φτάνουν στα δισεκατομμύρια που χάνονται από τους ε, κρατικούς κορβανάδες και που θα μπορούσαν να πάνε, πούμε, για διαφορέ πολιτικές, δημόσιε πολιτικές. Το θέμα είναι, λοιπόν, να μην χάνονται αυτά τα χρήματα, να μην τα, να μην τα χάνει ο προπολογισμό των κρατών μελών. Φυσικά υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρετε πολύ καλά ότι οι εγκληματίε όμω δεν σταματούν στα σύνορα. Είναι πολύ λογικό λοιπόν και εμεί να ανασκουμποθούμε. Και νομίζω ότι η ιδέα αυτή τη ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι η απαρχή αυτή τη διαδικασία, όπω είπε και η Επίτροπο πριν. Τώρα, σε 20 χρόνια, πώ θα διαμορφωθούν τα πράγματα, δεν μπορώ να το προβλέψω. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε επικοδομητικοί, θετικοί και να αρχίσουμε τέλο πάντων αυτή την προσπάθεια. Τα επόμενα πέντε χρόνια, ας πούμε, όταν ολοκληρωθεί αυτή η κοινοβουλευτική θητεία και η επόμενη, θα μπορούμε να έχουμε κάποια πράγματα από τα πετύχει. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και για τις πρακτικές δυσκολίες. Αλλά τέλος πάντων, πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα μιλήσω βουλγάρικα. Θα ήθελα να επευθύνω το πρώτο ερώτημα στον κύριο Μονάρ. Προτείνατε να προβούμε σε μία ανάλυση ή, εν πάση περιπτώσει, να λάβουμε υπόψη την αναλυτική συνιστόσα της Eurojust και της Europol, δηλαδή να δούμε ποιες είναι οι δραστηριότητες στα διάφορα κράτη-μέλη, μέχρι πού τα κράτη-μέλη μπορούν να ανταποκριθούν στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Αυτή η αυτός ο οργανισμός ή οι οργανισμοί πώς ε, ε, σχετίζονται με τα κράτη-μέλη και ποια είναι τα προσκόμματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πολυσχηδές αυτό φαινόμενο. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών και κρατών μελών. Δεύτερον, προς τον κύριο Μπάρνετ θα ήθελα να υποβάλω το εξής ερώτημα επιμείνατε ε, επί της χρήσης ε, των διαφόρων εξοπλισμών για τις υποκλοπές, ακροάσεις και για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Μπορείτε να μας πείτε πιο λεπτομερώς ποια είναι τα μέτρα που εφαρμόζεται για την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς. σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών. Δεν ήθελα να παρέμβω, αλλά θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια. Εγώ είμαι υπέρμαχος της επιχειρηματολογίας του κυρίου Μονάρ. Αφού άκουσα την Επίτροπο Ρέντινγκ, η οποία θέλει να προβάλλει μία πρόταση νομοθετικού περιεχομένου δυνάμει του άρθρου 86 για μία ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή περιορισμένης ευθύνης με δύο εναλλακτικέ ή την ομοφωνία που είναι πολύ δύσκολη ή την ενισχυμένη συνεργασία τον 9. Δηλαδή, ας το πούμε μια γενική εισαγγελία με... με τα δεκανίκια, με δεκανίκια για να μπορέσει να προχωρήσει. Συμμερίζομαι με τις ε, δυσκολίες που, τις δυσκολίες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτάσουμε σε υποδομές ασφάλειας. Υπάρχουν συνταγματικοί περιορισμοί στα κράτη-μέλη, καθώς και περιορισμοί από τις ίδιες τις ε, συνθήκες και ιδιαίτερα από την τελευταία, τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε. Η Ένωση δεν ολοκληρώνεται τάχιστα. Και αυτό αφορά και τις υποδομές ε, ασφάλειας. Θα ήθελα να τονίσω ότι στις υποδομές ασφαλείας δεν μπορούμε να αναθέσουμε περισσότερες αρμοδιότητες με λιγότερα μέσα. Όταν μιλάμε για τη Europol, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να πούμε σας δίνουμε νέες αρμοδιότητες για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο με 7 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Και δεν μπορεί να γίνει αυτό ενσωματώνοντας τη Europol και τις αρμοδιότητες της EpoL. Γι' αυτό συμφωνώ με αυτή τη λογική. Επίσης εκτιμώ ιδιαίτερα τα σχόλια και την εισήγηση του κυρίου Μπάρνετ, διότι Αυτά που συμβαίνουν σε μια τόσο ισχυρή ομοσπονδιακή χώρα, όπως είπα, αποτελούν μια εμπειρική συλλογιστική περί ασφάλειας. Γιατί υπάρχει σωρία οργανισμών στα πλαίσια της ασφάλειας, όμως αυτοί οι φορείς δεν ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα συνταγματικού δικαίου κάτι το οποίο είναι αδιανόητο για το δικό μας νομοθετικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσω για να ενισχύσω τις δύο παρεμβάσεις. Δηλαδή, για να τονίσω το, το ορθό της εισήγησης των δύο εισηγητών. Ο κύριος Μόναρ, για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω, απαντώντας στα σχόλια του κυρίου Νιούτον Ντάν, θεωρώ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ε, ένας από τους μεγαλύτερους συνεισφορείς για την ασφάλεια και εφαρμογή, εφαρμογή δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας εκλεκτός εταίρος της Europol και της Eurojust το ζήτημα είναι ότι μπορούμε να ε, έχουμε την πλήρη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου για αυτή την πολύ βασική συνεισφορά. Γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο του opt-out του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς τη συνεργασία του δικαστικού και δικαιοδοτικού τομέα, κάτι το οποίο θα ήταν ολέθριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας στην κυρία Βάιλερ, θα ήθελα να πω, δεν ήθελα να φανώ απεσιόδοξο, γιατί νομίζω ότι από τη δεκαετία του 90 έχουμε επιτύχει αρκετά στον τομέα της συνεργασίας αστυνομικών και διοκτικών αρχών σε θέματα δίωξης του εγκλήματος, αν λάβουμε υπόψη ότι έχουμε 27 κράτη-μέλη. Έχουμε δύο φορείς, δύο οργανισμούς. Μιλάμε για τη Eurojust και τη Europol που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο όλο εγχείρημα. Δεν υπήρχαν στην αρχή της ε, δεκαετίας του 90. Έχουμε μέσα, όπως το Ευρωπαϊκό Ένταλμα, ένταλμα Σύλληψης, κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο πριν από 20 χρόνια. Γι' αυτό έχει επιτελεστεί η πρόοδος. Απ' την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχουν ε, περιορισμοί που μας επιβάλλουν οι συνθήκες ως προς τις ε, αρμοδιότητες αυτών των οργανισμών και φορέων. Και υπάρχει και μεγάλη επιφυλακτικότητα από κράτη-μέλη να προχωρήσουν περαιτέρω. Γι' αυτό ε, υπάρχει ο κίνδυνος. Δεν λέω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή αποτελεί υπερφιλόδοξο σχέδιο. Αλλά αν κάνουμε ένα γιγάντιο βήμα προς τα εμπρός θα υπάρξει μεγάλη αντίσταση από το Συμβούλιο και έτσι θα χάσουμε αυτό το πολιτικό αρχικό κεφάλαιο το οποίο διαθέταμε. Δηλαδή πρόωρα προβάλλουμε πρωτοβουλίες πολλές φορές. Γι' αυτό μιλήσαμε και για την προοπτική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής για να ενισχύσουμε την Eurojust και τη Europol γιατί για να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή Χρειάζεται χρόνος. Αρχικά η εντολή θα είναι περιορισμένη και θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη και μόνο μερικά κράτη θα συμμετάσχουν. Δέχουμε λοιπόν μια παράλληλη στρατηγική. Ας ενισχύσουμε τους οργανισμούς που προϋπάρχουν χρηματικά και νομικά και μετά θα δούμε τι είναι δυνατόν από πλευράς Ευρωπαϊκής Αγγελικής Αρχής. Ως προς το δικό σας ερώτημα, κυρία Πρόεδρε, πώς μπορούμε να αποφύγουμε τους κινδύνους, γιατί η Γερμανία είναι η χώρα μου, είναι η πατρίδα μου και καταλαβαίνω τις δυσκολίες ενός ομοσπονδιακού συστήματος. Θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να ορίσουμε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ εθνικών αρχών και ευρωπαϊκών. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, η κυρία Ρέντινγκ μίλησε για 200 ε, συναντήσεις συντονισμού της ε, Eurojust τον τελευταίο χρόνο. Εδώ προσέρχονται ανώτεροι αξιωματούχοι, οι οποίοι κατανοούν ενδεχομένως καλύτερα τις προκλήσεις αυτές. Γίνεται ανταλλαγή απόψεων, υπάρχει διάδραση και θα κατανοήσουν το πλαίσιο καλύτερα. Αυτό είναι έμπρακτα ένας τρόπος επιτέλεσης πρόοδου και αυτό θα πρέπει να κάνουμε και σε καθημερινή βάση. Έτσι θα προετοιμάσουμε το έδαφος για ένα ευρύτερο ε, δικαιοδοτικό πλαίσιο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με ένα μόνο νομοθέτημα και δεν μπορεί να το δημιουργήσει μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν, να δίνουμε μια συνεχή όθηση και σε αυτό συνδράμει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη θετική του στάση εν γέννη. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Θα ξεκινήσω με το ερώτημα της Προέδρου. Ποιοι νόμοι και τεχνικοί χρησιμοποιήθηκαν για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Δεν θεωρώ ότι αυτό που κάναμε εμείς είναι λύση για όλους, αλλά στις Πολιτείες έχουμε το οργανωμένο έγκλημα υπό τη μορφή της μαφίας. Χρησιμοποίησαμε μυστικούς πράκτορες, υποκλοπές. Χρησιμοποίησαμε ειδικού νόμους δηλαδή, που μας το επέτρεπαν αυτό και Όλα αυτά είναι υπό την αιγίδα μιας ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Έχουμε την συγγελία που συνδέεται με τις διοκτικές αρχές που θα πρέπει να παρουσιάσουν σε έναν ουδέτερο δικαστή τα αποτελέσματα και θα, θα εκτιμήσει την ισχύ των αποτελεσμάτων υποκλοπών, θα δώσει κλητεύσεις και με μυστικές επιχειρήσεις ε, που επέτρεψε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για κάθε ομοσπονδιακή διοκτική αρχή, δηλαδή η κάθε ομοσπονδιακή διοκτική αρχή είχε το ρόλο της. Μετά το, την 11η Σεπτεμβρίου ε, κάναμε μεταρρυθμίσεις και είχαμε μια διαδικασία του α, ανώτατου δικαστηρίου, το Grand Jury. χρησιμοποιούμε αυτό το δικαστήριο για να διερευνήσει εγκλήματα στι ΗΠΑ ε, ήταν αποτελεσματικό, αποτελεσματική αυτή η προσέγγιση. Τώρα, για τις ε, συνταγματικέ δυσκολίες. Δεν θέλω εγώ να σας προτείνω μία λύση και όχι άλλη. Ο Ισπανός Ευρωβουλευτής μίλησε. Έχουμε διαφορές έχουμε όλοι μας διαφορές στο πώς οργανώνεται ας πούμε η εθνική αστυνομία στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ ας πούμε και σε όλο τον κόσμο. Ε, στην Αβία ε, μίλησα στην ε, αστυνομική ακαδημία, έδωσα μια ομιλία και μετά έκανα κάποιες συζητήσεις. Και κάτι που είναι γενικό κανόνα για την αστυνομία είναι ότι συχαίνεται το έγκλημα και θέλουν οι αστυνομικοί τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, υπάρχει μια καθολική κατανόηση των διαφορών, των δυσκολιών που έχουμε, των θεσμικών παραδόσεων κτλ. Κύριε Νιούτον Ντάν, ε, περιμένουμε να ταξιδέψει η Επιτροπή ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δούμε, να συζητήσουμε περισσότερο. Αλλά έτσι και εγωιστικά το βλέπω ως Αμερικανός. Ε, το θεωρούμε ευκαιρία το να μιλήσουμε για το διεθνές και διεθνικό έγκλημα, για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και με μεγάλη χαρά θα σας υποδεχτούμε στις ΗΠΑ. Ευχαριστώ τους ε, ομιλητές μας. Οι πληροφορίες που λάβουμε ήταν πολύ σημαντικές. Ε, είμαστε στην παραμονή της υιοθέτησης της βασικής έκθεσης της Επιτροπής ΚΡΙΜ. Πάμε τώρα ε, στο, στο τρίτο πάνελ με τίτλο «Προς ένα Ευρωπαίο Εισαγγελέα». Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Κούλα. Ελπίζω να τον προφέρω σωστά. Ο οποίος είναι τμηματάρχης ε, στην Όλαφ ασχολείται με θέματα ε, έρευνας και δίωξης των απατών. Η κυρία Κατλίν Λιτζέτη, επίκουρος καθηγητής ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, κανόνες για τις ποινικέ δίκες, ποινικέ διαδικασίες. Η κυρία Μισελ Κονίξ, πρόεδρος του Eurojust, ρόλος του Eurojust τη ε, για τη δημιουργία αυτού του, ε, της Ευρωπαϊκής ε, Εισαγγελικής Αρχής. Καλώς ήρθατε και οι τρεις. Nous la même Ίδια διαδικασία. Θα ακούσουμε καταρχάς τους τρεις ομιλητές. 15 λεπτά. Και συνεχεία θα τους ε, απευθύνετε ερωτήσεις. Euh, de, de dire votre, votre opinion. On va commencer avec uh, Monsieur Kuhl. Ο κύριος Κιόλ Ικούλ. Uh, ε, thank you. Uh... Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που δίνεται τον λόγο στην Όλαφ να παρουσιάσει την δική μας εξειδικευμένη ξεχωριστή εμπειρία με την διασύνδεση στην εντολή της ε, Επιτροπής ε, καθώς και σε σχέση με τη σχετική πείρα που υπάρχει για τον προβληματισμό αυτής της συγκυρίας για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως η κυρία Αντιπρόεδρος Επιτροπής, κυρία Ρέντινγκ, ήδη προανέφερε, η συνθήκη αναφέρει ως προτεραιότητα για την αρμοδιότητα του οργάνου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των απατών, της υπεξαίρεσης, της διαφθοράς και γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα να δούμε ποια είναι η δική μας πείρα που έχουμε συλλέξει με την εμπειρία μας ε, κατά τη διάρκεια αυτών των ετών λειτουργίας μας ε, στον αγώνα στη μάχη κατά της διαφθοράς ε, και του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προσπαθήσω με λίγα λόγια συνοπτικά να, να πω τι είναι εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει αυτά τα στοιχεία. Είναι προφανές για όλους ότι ιδιαίτερα σε σχέση με την οικονομική κρίση που διανύουμε σήμερα υπάρχει έντονη ανάγκη περαιτέρω να ενδυναμώσουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Αναφέρθηκε ήδη ότι υπάρχουν περικοπές ακόμα και για τα κονδύλια των αρχών αυτών που επιβάλλουν τον νόμο και διώκουν τους εγκληματίες και γι' αυτό πραγματικά αυτό παίρνει δραματικές διαστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι προφανώς πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο ξεπερνά τις δραστηριότητες ως διαχωριστικές γραμμές του οργανωμένου εγκλήματος και μάλιστα στην περίπτωση της Όλαφ μια μειοψηφία των περιπτώσεων δείχνουν και διασύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα. Αν δούμε όμως τα ποσά τα οποία εμπλέκονται, είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι συνειδητοποιεί κανείς αμέσως ότι το ίμιση των ποσών που διακυβεύονται είναι χρήματα που μπορεί κανείς ε, με μια πρώτη ματιά να δει μια τέτοια πιθανή διασύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα δηλαδή και αυτό δείχνει το, την εμβέλεια της απειλής ακόμα και αν είναι ένα περιορισμένο φάσμα ε, δραστηριοτήτων ε, αυτό το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουμε μπροστά μας σε σχέση με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, είναι απόλυτα λοιπόν σαφές ότι υπάρχει ανάγκη επίσης να δούμε και την πτυχή της εμπιστοσύνης που θα δείχνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και αυτό ξεκινά φυσικά με την εμπιστοσύνη που πρέπει να νιώθουν και να αισθάνονται οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο αυτό το θέμα. Πόσοι φορολογούμενοι θεωρούν ότι καλύπτονται και προστατεύονται τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δικά τους. Και εδώ πρέπει να το δούμε λοιπόν αυτό με βάση το βαθμό έκθεσης των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπονομεύονται από τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα και πρέπει να προστατευθούν. Αν δούμε τώρα τα γεγονότα ως από στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, πράγματι υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στη διάθεσή μας και είναι δυνατόν να ποσοστοποιήσει κανείς τουλάχιστον αυτά τα οποία υποβάλλονται από τα κράτη-μέλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια και αυτά τα οποία αναφέρονται ιδιαίτερα ως περιπτώσεις που με μια πρώτη ματιά μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει υποψία διάπραξης απάτης σε αυτές τις περιπτώσεις. Συλλέγονται αυτά τα στατιστικά στοιχεία όπως για παράδειγμα σε σχέση με τις πολιτικές του ε, Ταμείου Συνοχής, τις δραστηριότητες του Γεωργικού Ταμείου και μπορεί κανείς με βάση αυτά τα στατιστικά στοιχεία να ταυτοποιήσει και να εντοπίσει την έκθεση σε 500 εκατομμύρια ετήσια αυτού του ε, βαθμού ε, εμπλοκής και έκθεσης. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι είναι οι περιπτώσεις ε, αναφερόμενων απατών περιπτώσεων απατών που έχουν διαπιστώσει τα κράτη-μέλη και έχουν συνειδητοποιήσει ότι συμβαίνουν. Πρόκειται για περιπτώσεις απατών σε σχέση με άλλες μορφές τέτοιων περιπτώσεων ή υποψιών που μπορεί να έχουν τα κράτη-μέλη υποψιών για ατυπίες για παράδειγμα ή παρατυπίες. Τα μέσα και εργαλεία που η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει για τέτοιου είδους υποβολή τέτοιων στοιχείων, τέτοιων περιπτώσεων είναι τα μέσα και εργαλεία που χρησιμοποιούν οι διοικητικές αρχές των κρατών μελών και όχι οι αστυνομικές αρχές δίωξης. Οι περισσότερες λοιπόν από αυτές τις αρχές αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο ως ένα είδος παρατυπίας ε, χωρίς να διαπιστώνουν ή ανοιχνεύουν αν υπάρχει εγκληματική πρόθεση ή δόλος. Και οι περιπτώσεις αυτές είναι αρκετά υψηλότερες. Ο βαθμός ε, για παράδειγμα τέτοιων παρατυπιών είναι ανέρχεται σε ένα δίσα ετήσια. Και αυτό που μπορεί κανείς να πει είναι ότι πολλές φορές τα κράτη-μέλη απλά ικανοποιούνται με το να έχουν διαβιβάσει αυτά τα στοιχεία τέτοιων παρατυπιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει κάποια εξέταση, ε, ανάκριση περαιτέρω για την εγκληματική πρόθεση ειδόλο. Επαρκούνται σε αυτό. Ένα άλλο στοιχείο είναι το ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια από πλευράς δαπανών του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, γιατί έχουμε και το σκέλος των ιδίων πόρων. Και ήδη οι πόροι όχι μόνο καλύπτουν δασμού Τελωνιακού, αλλά επίσης και το τμήμα του ΦΠΑ, όσον αφορά αυτά που ε, εισπράττονται από τέτοια ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη. Και εδώ προφανώς η έκθεση σε δραστηριότητες ε, ε, οργανωμένου εγκλήματος, απάτες ε, δηλαδή κυκλικού χαρακτήρα, παίρνουν πολύ μεγάλες διαστάσεις. Υπάρχουν μελέτες που έχουν γίνει για αυτό το φαινόμενο και αληθεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μικρότερο τμήμα στην ίσπραξη του ΦΠΑ σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Όμως, αν εξετάζουμε τη δυνατότητα της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προφανώς και αυτή αυτή η διάσταση, αυτή η συνιστόσα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όσον αφορά διασυνοριακά την ίσπραξη ΦΠΑ. ΦΠΑ που εισπράτεται μέσα στο πλαίσιο για παράδειγμα προϊόντων μαρμούδων απομίμησης που εισάγονται με τέτοιες περιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να καταπολεμηθούν. Μια άλλη πτυχή επίσης είναι ότι πρέπει τα δικήματα διαφθοράς να δει κανεί ότι υπονομεύουν και αυτά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο που είναι δύσκολο, είναι δυσχερέστερο να ποσοστοποιηθούν, να υπολογίσει κανείς την πραγματική διάσταση αυτής της ε, ζημιάς που υφίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτές τις περιπτώσεις. Ποια είναι η κατάσταση που έχουμε μπροστά μας. Χαρακτηρίζεται από αρμοδιότητες ε, διοκτικές ε, και ε, ποινικού δικαίου από πλευράς των κρατών μελών και η Όλαφ συνεργάζεται, συνεργαζόμενη με αυτές τις αρχές των κρατών μελών είδαμε ότι τα τελευταία 12 χρόνια από τη δημιουργία, τη συγκρότηση της Όλαφ ότι καταφέραμε πετύχαμε πολλές ιστορίες επιτυχίας, με επιτυχή έκβαση, περιπτώσεις που με επιτυχή τρόπο ε, διαφωτίστηκαν και ε, ε, έδειξαν το τι ακριβώς συμβαίνει. Επίσης και σημαντικές κυρώσεις ως ποινές επιβλήθηκαν κατά τα τελευταία 12 χρόνια. Για παράδειγμα 900 έτη φυλάκισης που επευλήθησαν ως ποινές στους εγκληματίες υπεύθυνους το γεγονός όμως είναι ότι με την δικαστική αρχή υπάρχουν βραδύτεροι ρυθμοί, μάλιστα ιδιαίτερα βραδείς ρυθμοί ε, δράσης και κινητοποίησης. Σε διαφορετικό θα έλεγα, σε διαφορετική ένταση έχουμε και σε σχέση με την ε, περίπτωση περιπτώσεων που διαβιβάζονται από τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλές οι οποίες μια και βασίζονται σε σχέση και με τα στοιχεία που συντάσσονται από την ίδια την Όλαφα με τα τεκμήρια και τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί και αξιολογηθεί από την Όλαφ πρέπει να δούμε ότι στο επίπεδο της δικαστικής δίωξης έχουμε διαφοροποίηση σε σχέση με τις αθωτικές αποφάσεις δικαστηρίων που και αυτές λαμβάνουν χώρα και πρέπει να δούμε με το αντίστοιχο άρθρο ότι η καταπολέμηση των απατών πρέπει όμως να στέφεται με επιτυχία, πρέπει να είναι αποτελεσματική, πρέπει να είναι πιστική και αποτρεπτική και δεδομένη της κατάστασης με τις αθωτικές αυτές αποφάσεις ε, και την διαρροή, α το πω έτσι, διαφυγή ε, των υπευθύνων είναι αμφισβητήσιμο αν είμαστε τόσο αποτελεσματικοί και βλέπουμε ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό αυτών των περιπτώσεων περίπου 50 κιόλας μπορεί κανείς να πει τις 100 από αυτές τις περιπτώσεις δεν οδήγησαν σε καμιά καταδίκη από πλευράς δικαστηρίων των υπευθύνων που θα έπρεπε να είχαν καταδικαστεί. 50% περίπου είναι το ποσοστό των δράσεων που καταλήγουν από τα κράτη-μέλη σε τέτοιες, ε, ε, ας το πω έτσι, ακυρώσεις δικών ή μη συνέχεια στην δικαστική δίωξη. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Έχουμε σε κάποια κράτη-μέλη 90% καταδικαστικές αποφάσεις σε σχέση με όσες περιπτώσεις καταλήγουν στα δικαστήρια, σε άλλες περιπτώσεις μόνο 20 όμως 100. Τι δείχνουν αυτά τα διαφορετικά μεταξύ τους στοιχεία. Δείχνουν ότι υπάρχει έντονη ανάγκη να βελτιωθεί περαιτέρω το σύστημα, ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικό και περισσότερο συνεκτικό αναλογικά, πιο ε, αποτελεσματικό. Ένα άλλο στοιχείο είναι η διασυνοριακή, διακρατική διάσταση σε σχέση με τα όσα εξετάζονται και αυτό στενά συνδέεται με τον χαρακτήρα αυτών των περιπτώσεων που είναι περιπτώσεις που σχετίζονται με τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά π.χ. προϊόντα τα οποία έχουν μέσω λαθεμπορίου εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαμετακομίζονται μεταξύ διαφορετικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από, το, από ένα σε άλλο. Ακόμα και με τέτοιου είδους δαπάνες έχουμε δαπάνες που εγκρίνονται μόνο υπό τον όρο ότι κάποια, ε, κάποιο τέτοιο πρόγραμμα ή σχέδιο έχει διασυνοριακό χαρακτήρα και αυτό πάλι δημιουργεί συγκεκριμένες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν όσον αφορά τις ε, διακριβώσεις και ανακρίσεις από πλευράς των κρατών μελών υπάρχει κατάτμιση και πολλές φορές κατακαιρματισμός και περιορίζεται πολλές φορές ο χρόνος ε, για την προσαγωγή τέτοιων, ε, αυτών των υπευθύνων, των υπευθύνων τέτοιων αδικημάτων στα δικαστήρια. Έχουμε και αρνητικές περιπτώσεις ε, σε σχέση με τις σχέσεις των δικαστικών αρχών ή μεταξύ των διοκτικών αρχών όπου καμιά από αυτές τις αρχές δεν δέχεται να οδηγήσει στα δικαστήρια αυτή την περίπτωση ισχυριζόμενη λέγοντας ότι υπάρχει τέτοια, τέτοια πολυμορφία μεταξύ των των τεκμηρίων που δεν είναι δυνατόν να αποφασιστεί πού ακριβώς μπορεί να εκδικαστεί μια τέτοια υπόθεση, ποιος θα ήταν τελικά αρμόδιος. Και μεταξύ τέτοιων αντικρουωμένων περιπτώσεων είναι πολλές φορές δύσκολο οι εθνικές αρχές να δώσουν συνέχεια σε μια τέτοια περίπτωση δίωξης και να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν ε, με υψηλότερο βαθμό προτεραιότητας από ό,τι συνήθως ε, αντιμετωπίζονται τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό δείχνει ότι σε σχέση με αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ανάγκη να ε, υποστηρίζονται από τεχνική πραγματογνωμοσύνη. Πρέπει να υπάρχει πολύ καλή κατανόηση των ευρωπαϊκών κανονισμών και διατάξεων που ισχύουν και πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε σχέση με τη διάθεση ευρωπαϊκών κονδυλίων αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Περιορίζονται κάποιες αρμοδιότητες σε σχέση με τις δυνατότητες διοκτικών σωμάτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχει όμως διακριβωτική, ανακριτική ή διοκτική αρμοδιότητα με σαφή τρόπο που να μπορεί να δίνει συνέχεια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αν θέλουμε και θα θέλαμε να είχαμε πρόσβαση σε συγκεκριμένες ε, πληροφορίες στον τραπεζικό τομέα για παράδειγμα είναι αδύνατο, είναι ανέφικτο η Όλαφ να συλλέξει όλα αυτά τα στοιχεία τραπεζικού χαρακτήρα Μπορεί κανείς να προσπαθήσει να διακριβώσει ποιος είναι εκείνος ο οποίος επωφελείται από κάποια κεφάλαια. Όταν έχουμε όμως το θέμα της ε, εξακρίβωσης αν κάποια τραπεζικά τέτοια στοιχεία είναι αξιόπιστα και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι, δημιουργούνται πολλές δυσχέρειες. Και σε σχέση με το μέσο, το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως προανέφερε η κυρία Ρέντινγκ, θα πρέπει ανεξάρτητα να μπορεί να δρά πανευρωπαϊκά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να έχει μια μια τέτοια διοργανωτική δομή ώστε να μπορεί να εντάσει τις εθνικές αρχές σε αυτήν και η ίδια να μπορεί να λειτουργεί μέσω αυτών αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει και ένα τμήμα δίωξης και διακριβώσεων που θα μπορεί να ε, οδηγεί, να καθοδηγεί τις ανακριτικές και διοκτικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη και να έχει μια πλήρη επισκόπηση ε, συνολικά του τι συμβαίνει και πώς ε, δίνεται συνέχεια σε κάποια υπόθεση. Και όλα αυτά επίσης με το να τονίσουμε ότι αυτά θα πρέπει να βασίζονται στους υφιστάμενους πόρους και δυνατότητες. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τους διαθέσιμους πόρους ε, με το πιο αποτελεσματικό τρόπο μέσω, όλα, μέσω της Eurojust, της Europol, ώστε να μπορέσουν όλα αυτά να συγχωνευτούν και να συγκλίνουν στην καλή λειτουργία ενός ευρωπαϊκού εισαγγελικού τέτοιου θεσμού ως μέσου. Αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε και καλύτερα αποτελεσματικότητα. Καλύτερη αποτελεσματικότητα ώστε να καταδικάζονται, να προσάγονται στα δικαστήρια και να καταδικάζονται ε, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό οι υπεύθυνοι από ό,τι σήμερα, από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Είναι αυτά όλα πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Δεύτερον, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όπως όλοι όλοι γνωρίζουν λειτουργεί, λειτουργεί μέσω συγκεκριμένων πιλωτικών τομέων και δράσεων όπου συγκεκριμένα συλλέγεται πείρα και έχουμε ήδη συγκεκριμένη πείρα σε αυτούς τους τομείς. Χρειαζόμαστε σαφώς την υποστήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν χρειάζεται. Νομίζω περιτεύει να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το εγχείρημα ποτέ δεν θα είχε καμία πιθανότητα να ευδοκιμήσει μέσω της συντακτικής συνέλευσης, μέσω δηλαδή τελικά της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, αν δεν υπήρχε η στεναρή υποστήριξη και βούληση των Ευρωβουλευτών. Και ήταν το Ευρωκοινοβούλιο εκείνο το οποίο έδωσε εντολή να συνταθούν μελέτες, όπως για παράδειγμα για το όργανο, για το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όλα αυτά είναι πράγματα στα οποία θα έπρεπε να εμπλέκεται πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να διαδραματίζει από αυτόν ένα πολύ ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο. Αποκινούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Uh, and now, Mrs. Uh, ευχαριστώ, κυρία Λιγκέτη. Members of uh, Parliament. Um... Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να αναφερθώ μόνο σε ένα ζήτημα. Είμαι πεπισμένη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή χρειάζεται κανόνες που να βασίζονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο με βάση τις διοκτικές αρχές και αρμοδιότητες ανακριτικές και διοκτικές. Διαφορετικά θα μιλάμε για Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, αλλά δεν θα είναι μια τέτοια αρχή. Πριν μιλήσω για τα επιχειρήματά μου, για να υποστηρίξω την εισήγησή μου αυτή, θα ήθελα να μιλήσω για τη συνθήκη. Το άρθρο 86 ορίζει πολύ σαφώς ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα είναι υπεύθυνη για την ε, ανάκριση, δίωξη και καταδίκη των εγκληματικών στοιχείων. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα είναι άμεσα υπεύθυνη για την ανακριτική φάση και τη δίωξη. Και πολλοί μίλησαν για τη διατύπωση της συνθήκης τι σημαίνει από πλευράς της ε, Eurojust. Αν διαβάσουμε το άρθρο 86, καθίσταται σαφές ότι δεν μπορούμε παρά να έχουμε ένα όργανο το οποίο να έχει δικαιοδοτική ισχύ για ανάκριση και δίωξη ε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Αλλά αυτό το σχήμα δεν μπορεί να είναι πάντα λειτουργικό. Δυνάμει λοιπόν του άρθρου 86 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα πρέπει να είναι άμεσα υπεύθυνη αυτή της διαδικασίας ε, ανάκρισης και δίωξης του εγκλήματος. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσω για αυτό τον ε, συσχετισμό μεταξύ Eurojust και EPPO γιατί έγινε λόγος για το διεθνές, για την διεθνή εγκληματικότητα. Το άρθρο 86 δεν αναφέρεται στο διεθνές έγκλημα, σε αυτή τη διεθνή διάσταση του εγκλήματος. Και με βάση τα στοιχεία και τα επιχειρήματα του κυρίου Κούλ, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να περιοριστούν οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αγγελικής Αρχής ε, ως προς τη δίωξη του διεθνούς εγκλήματος. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη το, τη συνιστόσα της συνεργασίας με τη Eurojust. Η Ευρωπαϊκή Αγγελική Αρχή θέλει να υπερβεί αυτή τη διάσταση και να ανακρίνει, να διώκει και σε μεμονωμένα σε ένα κράτος μέλος. Αλλά μία τέτοια διοκτική αρχή δεν μπορεί να είναι παρά μία ενιαία δικαιοδοτική αρχή. Παρά το γεγονός ότι πλήττεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εμπλέκονται σε αυτά τα ε, υποτιθέμενα αδικήματα, και θα πρέπει να υπάρχει ενιαία προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη στιγμή που πλήττονται περισσότερες από μία δικαιοδοσίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή δεν μπορεί να ε, παρέμβει, διότι ε, εδώ μιλάμε για τον διεθνικό χαρακτήρα του εγκλήματος. Η κυρία Ρέντιν μας είπε σήμερα το απόγευμα ότι η Επιτροπή θα προβάλλει μια πρόταση για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής που βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο αλλά αποκεντρωμένο πρότυπο. Η Επίτροπος σιώπησε ως προς το διαδικαστικό σκέλος το οποίο όμως είναι ζωτική σημασίας για αυτό το ολοκληρωμένο αλλά και αποκεντρωμένο σχήμα. Είναι αυταπόδεικτο ότι όσο πιο αποκεντρωμένο είναι το πρότυπο, τόσο περισσότερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα εθνικά δικαιοδοτικά συστήματα και όσο πιο συγκεντρωτικό, τόσο περισσότερο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ευρωπαϊκή του διάσταση εκ προημίου. Αυτό το ολοκληρωμένο και αποκεντρωμένο πρότυπο δεν ορίζει εκ των προτέρων ε, ποιο διαδικαστικό σχήμα θα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκείνοι που εκπονούν τα πολιτικά σχήματα θα πρέπει να το σκεφτούν αυτό πιο σοβαρά. Μπορούμε να προβλέψουμε λοιπόν αυτό το ολοκληρωμένο και αποκεντρωμένο σύστημα με βάση το εθνικό δίκαιο, όπου η αποκεντρωμένη εισαγγελική αρχή θα δίνει εντολές στις εθνικές ανακριτικές αρχές και εισαγγελικές αρχές με βάση το ε, υπάρχον δίκαιο. Αυτή η αποκεντρωμένη εισαγγελική αρχή θα συνεργαστεί με τους εναρμονισμένους ε, κοινοτικούς ευρωπαϊκούς νόμους και είμαι υπέρ αυτής της δεύτερης εναλλακτικής για τρεις λόγους. δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το εθνικό πρότυπο δικαίου, διότι η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής εισαγγελική Αρχής θα ήταν ε, θύμα μεταβλητής γεωμετρίας. Σήμερα το απόγευμα μιλήσαμε για διαφορετικά δικαιοδοτικά συστήματα και διαδικαστικά στα κράτη-μέλη. Εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή έχει ανακριτικό και διοκτικό χαρακτήρα με βάση τα εθνικά δίκαια, σημαίνει ότι οι εξουσίες της εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη με στα πλαίσια της ανάκρισης και δίωξης. Ε, ε, εάν πρέπει να γίνει έρευνα κατοίκων, για παράδειγμα, σε ένα κράτος χρειάζεται ε, μια εισαγγελική εντολή για να διενεργηθεί μια έρευνα κατοίκων. Σε άλλα κράτη-μέλη, ο, ο εισαγγελέα ο ίδιος μπορεί να δώσει, να διοδοτήσει για κάτι τέτοιο. Εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή βασιστεί στο εθνικό ποινικό δίκαιο, είναι σαφές ότι θα επαφίεται στη χώρα όπου γίνεται η δίωξη, η έρευνα. Πολλές φορές δεν χρειάζεται η εισαγγελική εντολή άλλες χρειάζεται. Εκεί που δεν χρειάζεται έχει περισσότερη δικαιοδοσία. Αυτές οι διαφορές εξουσιών θα οδηγούσαν σε ένα τύπο forum shopping και αυτό θα ήταν επιζήμιο και για τον κατηγορούμενο. Νομίζω λοιπόν ότι όταν βασιζόμαστε στο εθνικό ποινικό δίκαιο, τότε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα είναι θύμα των εθνικών αρχών. Και σε αυτή την ε, περίπτωση θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούν να προβληθούν κατεξιοδότηση πράξεις. Θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα και θα επανέλθω στις συστάσεις ή τα παραδείγματα που μας έδωσε και ο κύριος Μπάρνετ. Μας είπε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος, με βάση τη δική του πείρα, στη ΣΥΠΑ, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος χρήσης πρακτόρων υποκάλυψη ή υποκλοπών για το οργανωμένο έγκλημα ε, αφορά παρεμβατική ανάκριση ή έρευνα και δεν ρυθμίζεται κατά τον ίδιο τρόπο από τα διάφορα κράτη-μέλη. Για να επανέλθω στις ε, υποκλοπές, ξέρετε ίσως ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπονται αλλά δεν μπορούν να προβληθούν ως αποδεικτικό στοιχείο ε, στο δικαστήριο, απλώς ως εφαλτήριο για να συλλεγούν περισσότερα στοιχεία. Επίσης, τα οπτικοακουστικά ε, αυτά μέσα απαγορεύονται σε, σε μια χώρα όπως την Ισπανία, ενώ επιτρέπονται σε άλλες 26. Η επιγραμμική, η online ε, έρευνα δεν επιτρέπονται στο Λουξεμβούργο ε, και στην Ολλανδία. Απαγορεύονται και στην Ιταλία και στην Πολωνία, ενώ σε άλλες χώρες θεωρείται ένα σύνομο ανακριτικό μέσο. Αυτές οι διαφορές με βάση τον εθνικό νόμο θα σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα έχει ευρύτερες εξουσίες στα κράτη Α και πολύ πιο ε, συσταλτικά μέσα όταν ερευνά σε άλλα κράτη. Θα πρέπει λοιπόν να μην σταθεί αυτό επισήμιο και για τον εναγόμενο, ιδιαίτερα γιατί και εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρετε μεγάλη ευθύνη. Έχετε ε, προβάλει πολλά μέτρα και συστάσεις ως προς τις ρήτρες διασφάλισης, διαδικαστικές ρήτρες διασφάλισης και Αυτές οι διαφορές θα ήταν επιζήμιες ε, ως προς τη διασφάλιση των συμφερόντων. Έμπρακτα, ο εναγόμενος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα δίκαιας δίκης, κάτι το οποίο δεν θα μπορεί να γίνει τη στιγμή που ισχύει διαφορετικός νόμος μέσα στα πλαίσια της ανάκρισης και δίωξης, διότι ο εθνικός νόμος ισχύει επιμεριστικά και αυτό αφορά και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του εναγόμενου. Άρα η εισαγγελική αρχή δεν μπορεί να διασφαλίσει τα δικαιώματα του εναγόμενου και ο εναγόμενος δεν θα μπορεί να κατανοήσει ποιες ρήτρες διασφάλισης ισχύουν με βάση την ανακριτική διοκτική διαδικασία στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και συνεπώς πώς ε, θα στερείται του δικαιώματος παροχής δίκαιας δίκης με βάση τα άρθρα 5 και 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γι' αυτό θα ήθελα να υποστηρίξετε την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Εάν φτάσει στο δικό σας τραπέζι, θα πρέπει να μιλήσετε για ενιαίους κανόνες εφαρμογής σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ, κυρία Λιγκέτη. Και τώρα έχουμε τελευταία παρουσίαση. Την κυρία Μισελ Κονίξ, πρόεδρου της Eurojust, για το ρόλο της Eurojust κατά τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Γραφείου Εισαγγελέα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτές. Με μεγάλη χαρά μπορώ να σας πω κάποια στοιχεία για το πώς ε, εργάστηκε μέχρι τώρα το Eurojust και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος του αν δημιουργηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έποθα τη λέω από εδώ και στο εξή. Πριν από 12 χρόνια αρχίσαμε να δουλεύουμε εδώ στις Βρυξέλλες 15 άτομα, πολύ θετικά το βλέπαμε και πιστεύαμε ότι τα κράτη-μέλη ήταν ε, σε θέση να καταπολεμήσουν το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, αλλά πιστεύαμε επίσης ότι θα μας εμπιστευόταν έναν ειδικό ρόλο ε, για να τους διευκολύνουμε, για να συντονίσουμε τη δουλειά μας, για να καταπολεμήσουμε αυτό το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα. Το βλέπαμε αισιόδοξα, παρά το γεγονός ότι κάποιες δικαστικές αρχές ε, σε κάποια κράτη-μέλη ε, λέγανε ότι αυτό είναι επιστημονική φαντασία στον χώρο της νομικής, της δικαιοσύνης. 12 χρόνια μετά, η Eurojust είναι Πραγματικό φορέας, υπάρχει συντονισμός, υπάρχει συνεργασία, ενισχύουμε τον αγώνα κατά του σοβαρού ε, διοργα... διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματο. και μέσω αυτής της συνεργασίας είμαστε μοναδικοί στον κόσμο. Πουθενά δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο με εμάς. Ούτε στην Νότια Αμερική, ούτε στον Αραβικό κόσμο δεν υπάρχει το Arab Just και, και ούτω καθεξής. Εμείς το κάνουμε σε αυτόν τον αγώνα κατά πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Όταν βλέπετε τα νούμερα, βλέπετε ότι από το 2002 μέχρι το 2012 κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των κρατών μελών, σιγά σιγά χτυπούσαν όλο και περισσότερο στις πόρτες μας και πέρυσι είχαμε 1532 υποθέσεις. Ενώ όταν ξεκινήσαμε είχαμε 200 υποθέσεις. Βλέπετε λοιπόν την τρομερή διαφορά. Τώρα, να προχωρήσουμε και αν κοιτάξουμε τι υποθέσεις αντιμετωπίζουμε. Τα πρώτα 10 χρόνια είχαμε το λαθρεμπόριο εργών ναρκωτικών, απάτη και εξέπλυμα χρήματος. Και πέρυσι Η απάτη είναι πιο σημαντική από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Και τώρα έχουμε την απάτη, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών με αυτή τη σειρά και το οργανωμένο έγκλημα, τρίτο. Επίσης, λίγες υποθέσεις έχουμε για τη διαφθορά και τα εγκλήματα εναντίον των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απάτη, Όμω είναι εντυπωσιακό τμήμα τη καθημερινή δουλειά μα. Όλε οι μορφέ απάτης. ΦΠΑ, ε, η απάτη καρουσέλ. Παραδείγματος χάρη απάτη στα φρούτα και τα κρέατα. Καθημερινά έχουμε τέτοιε υποθέσει. Όλα αυτά μεταφράζονται σε χρήματα. Γιατί όλε αυτέ οι απάτες γίνονται για το χρήμα. Όπως είπα, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών επί πολλά χρόνια ήταν ε, οι περισσότερες υποθέσεις. Είχαμε κατασχέσεις κοκαίνης, ε, ναρκωτικών. Ε. Και οι εγκληματίες λαθρεμπόριο ναρκωτικών αγόραζαν και ακίνητα με αυτά τα λεφτά. Στη Σουηδία το Μάρτιο, μετά από δύο χρόνια συντονιστικών προσπαθειών, καταφέραμε να διώξουμε επιτυχώς και πάνω από 14 συντονιστικές συναντήσεις καταφέραμε να τους καταδικάσουμε και να δημεύσουμε τα προϊόντα του εγκλήματος. Επομένως, η, δικαστική συνεργασία, η αποτελεσματική δικαστική συνεργασία οδηγεί σε αποτελέσματα. Η συνθήκη της Λισαβόνας, το άρθρο 86, λέει ότι υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσουμε ε, μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γραφείο. Ευχαριστώ. Και μπορούμε να καταπολεμήσουμε τα εγκλήματα που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας θα είναι υπεύθυνο για την έρευνα, δίωξη και εκδίκαση. Πέρα από τη διευκόλυνση λοιπόν των δικαστικών αρχών για την ε, έρευνα και δίωξη, αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι το ΕΠΟ θα πρέπει να εξασφαλίσει και την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών. Χρειάζεται όμως ομοφωνία. Αν δεν επιτευχθεί υπάρχει η ενισχυμένη ε, συνεργασία με τη συμμετοχή εννέα ευρωπαϊκών χωρών, εφόσον, αυτές, εφόσον εννέα χώρες ε, συμφωνήσουν. Τώρα, η ΕΠΟ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως νέος παίχτης. Χαρακτηριστικά για να λειτουργήσει το σχήμα. Θα πρέπει να ενταχθεί στο σημερινό πλαίσιο της ε, αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας. το είπαμε, όλα το απόγευμα το λέγαμε. Μέσα σε εποχή οικονομικής λιτότητας, όπου δεν πρέπει να ξοδεύουμε, θα πρέπει κάθε δραχμούλα, κάθε δεκάρα να την προστατεύουμε. Κάθε σέντ, κάθε ευρώ. Και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά το σύστημα. Που προβλέπει αστυνομική και δικαστική συνεργασία βέβαια. Επίσης, πρέπει να υπάρχει στενή σχέση με τις αρμόδιες εθνικές αρχές αρχές που ε, ερευνούν τέτοιες υποθέσεις σε εθνικό επίπεδο και σχέση του ΕΠΟ με τα δικαστήρια των κρατών μελών, για να δούμε τα δικαιοδιωτικά θέματα. Γιατί στο βαθμό που δεν θα υπάρχουν τέτοια ευρωπαϊκά δικαστήρια, θα πρέπει η Εθνική Εισαγγελής να εκδικα... να προσκομίζουν στο δικαστήριο υποθέσεις που έχει διερευνήσει το ΕΠΟ. Αλλά σε ποιο δικαστήριο, στα δικά του εθνικά δικαστήρια. Ε, θα πρέπει λοιπόν όλοι οι φορείς να συνεργαστούν, να συντονιστούν και για να είναι αποτελεσματικοί θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι με την Europol και την Όλαφ να βασιστούμε στην εμπειρία, στην πραγματογνωμοσύνη, στη γνώση και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε συνέργειες όπου αυτό είναι δυνατό. I send out today a strong message. Ένα ισχυρό μήνυμα θέλουμε να απευθύνουμε σήμερα, διότι όλα αυτά τα χρόνια συνεισφέρουμε για την ανάπτυξη αυτών των θεμάτων. Έχουμε εμπλακεί στον προβληματισμό και προβληματιστήκαμε επί μεγάλο χρονικό διάστημα πώς μπορεί κανείς να συνεισφέρει και τι μπορεί να κάνει κανείς. Ό,τι και να κάνει κανείς πρέπει να το κάνει παράλληλα με την Eurojust. Και γιατί αυτό, διότι βλέπουμε ότι σε περίπτωση αυτής της ε, δυνατότητας θα πρέπει με διευρυμένη συνεργασία να μπορέσουμε να δράσουμε και να προχωρήσουμε. Αυτό είναι κάτι που με βεβαιότητα μπορούμε σήμερα να το πούμε. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα είναι αναγκαίο συντονιστής η Eurojust που θα πρέπει να σε σχέση με τα συμμετέχοντα και μη συμμετέχοντα κράτη-μέλη να διασφαλίζει αυτή την τροχή, αυτή την πορεία. Και κάτι άλλο το οποίο γνωρίζαμε και προηγούμενα δηλαδή για τις παραβιάσεις ε, και παραβάσεις εις βάρος των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διασύνδεση με περιπτώσεις ε, οργανωμένου εγκλήματος θα πρέπει η Eurojust σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ε, δράσης να μπορεί να εμπλέκεται και να δρά και θα συντονίζει τις δράσεις του EPPO και των, τις δράσεις των εθνικών αρχών σε αυτό το πλαίσιο. Αυτά τα δύο πράγματα τα γνωρίζουμε με βεβαιότητα ήδη τώρα. Διευρυμένη συνεργασία που αυτή θα λειτουργήσει στις περισσότερες περιπτώσεις και η ανάγκη διασφάλισης του συντονισμού με τα παράλληλα συνδεόμενα εγκλήματα. Τι άλλο θα μπορούσε να προσθέσει κανείς. Η πρόσθετη αξία είναι το στοιχείο που θα μπορούσε να αναφέρει κανείς σε σχέση με την συνεργασία και συντονισμό με τρίτες χώρες. Και αυτό αληθεύει σε σχέση με τις περιπτώσεις που εξετάζαμε και αντιμετωπίσαμε πολύ συχνά μας οδηγούσαν και βρεθήκαμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν εδώ η ανάγκη να συνεργαζόμαστε με τρίτες χώρες σε αυτά τα πλαίσια. Επίσης να υπάρχει διασύνδεση και συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές των κρατών μελών είναι προφανές ότι οι διοκτικές δράσεις, ε, η διοξική από πλευρά ε, δικαστικών αρχών πρέπει να διασφαλίζεται στο επίπεδο των κρατών μελών. Χρειάζονται σαφείς διασυνδέσεις λοιπόν και συνεργασία με αυτές τις κρατικές αρχές αυτών των κρατικών αρχών. Στη Eurojust επικεντρωθήκαμε μέχρι σήμερα με ιδιαίτερο τρόπο και έντονα στη διασφάλιση αυτών των κομβικών σημείων και συνεργασίας μεταξύ Eurojust και των εθνικών συντονιστικών συστημάτων των κρατών μελών και αυτό είναι θέμα κάθε κράτους μέλους, να διασφαλίζει αυτή τη διασύνδεση με τις περιπτώσεις που εξετάζονται στο κράτος μέλος αυτό και τις ίδιας της δράσης της Eurojust. Συντονιστικά υπάρχουν μέσα και εργαλεία και έχουμε και την ε, περίπτωση από πλευράς Eurojust ε, με την ανταλλαγή πληροφοριών από και προς ε, τα κράτη-μέλη, από και προς την Eurojust. Τι άλλο μπορούμε να πούμε. Έχουμε και σχέσεις συνεργασίας και με την ε, Europol και με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και όλα αυτά από πλευράς του καθηγητού Μονά σε σχέση με την Europol και με την ε, διασύνδεση με τα εστιακά κέντρα για την ανάλυση και αξιολόγηση 80% αυτών των κέντρων εστίασης ε, με την δυνατότητα διασφάλισης, διασύνδεσης ε, με την ε, Europol και με την Όλαφ επίσης έχουμε διασφαλίσει ασφαλή διασύνδεση και πέρυσι και διασφαλίσαμε ότι θα εμπλέκεται η ώρα, θα εμπλέκεται σε πέντε τέτοιες περιπτώσεις ε, για τον συντονισμό και την δίωξη. Και η γραμματεία που υφίσταται επίσης και στη Eurojust και σε κάποιες από τις εθνικές αρχές και κομβικές, ε, ε, κομβικά τέτοια σημεία της Eurojust σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Υπάρχει και αυτή η ας το πω έτσι ε, εγκύτητα με την Europol και σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μέσα από το EPPO σε ένα κύκλο ζωής ή δράσης μέσα σε τρεις φάσεις. Η αναφορά σε σχέση με τις υποψίες που υπάρχουν υπόπτων, υπόπτων περιπτώσεων, η ΕΠΠΟ που θα αποφασίζει αν θα ανοίξει κάποια δράση ε, ανακριτική ή άλλη. Επίσης ε, οι, δίο οι διοκτικές δράσεις που αποφασίζονται ή ε, αρχίζουν να δρομολογούνται και βλέπουμε έτσι ότι υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης στο τέλος τέλος ε, των αποφάσεων, δηλαδή προσαγωγή στα δικαστήρια, δικαστική απόφαση και εκτέλεση της απόφασης. Σε κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά πρέπει να διασφαλίζουμε τη συνέχεια και την ολοκλήρωση. Και η Eurojust θα μπορούσε να έχει να, έχει, να ολοκληρώνει και να αντανακλά αυτές τις ε, δράσεις, αυτούς τους κύκλους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να βασίζεται σε μια δυνατότητα διευρυμένης συνεργασίας απαραίτητο ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει με έτσι με αυτή τη δράση της είτε μέσα στο πλαίσιο της συναπόφασης που προβλέπεται σε σχέση με αυτές τις δράσεις από πλευράς Eurojust ή για το πώς η Eurojust με βάση το άρθρο 85 θα μπορεί να δρά με επαυξημένες δραστηριότητες και καθήκοντα σε όλες αυτές τις επιμέρους φάσεις βλέπουμε ότι η Eurojust θα μπορούσε, θα μπορεί να διαδραματίζει ένα σπουδαίο ρόλο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν όλα να καταστούν σαφέστερα με την επικέντρωση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα είμαι σύντομη σε σχέση με αυτές. Είναι περιπτώσεις ε, που βασίζονται σε σχέση με πραγματικά γεγονότα. Για παράδειγμα, μια ισπανική εταιρεία με ε, συμφέροντα σε, διαφορετικά, σε διαφορετικούς τομείς, ε, γεωργία, πετρέλαια, τρόφιμα και για παράδειγμα βλέπουμε ότι γίνονται ε, αναλαμβάνεται ε, δράση ανακριτική σε σχέση με αυτές τις διαφορετικές πτυχές και θα αποφασιστεί στη συνέχεια η δίωξη. Υπήρξε καταδίκη για την δικτύωση μέσω εταιριών σε σχέση με τον Παναμά, τις ε, κάτω χώρες ε, και την ε, δυνατότητα πολυεθνικής δράσης. Αν υποθέσουμε ότι με βάση τις δράσεις της Eurojust διαπιστώνεται ότι η φοροδιαφυγή και τα συναφή μπορούν να οδηγήσουν στην τεκμηρίωση ευρωπαϊκού χαρακτήρα απάτησης βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαπιστώνεται ότι στην Ισπανία συνέβησαν αυτές οι εγκληματικές πράξεις και στο Βέλγιο. Υποθέτοντας τώρα ως υπόθεση εργασίας ότι η Ισπανία και το Βέλγιο είναι δύο χώρες που συναπαρτίζουν μεταξύ τους και αποτελούν κράτη-μέλη της EPPO, ε, τότε η Eurojust θα πρέπει να ε, ζητήσει σε μια συντονιστική, συντονιστικού χαρακτήρα δράση από πλευράς των κρατών μελών να οδηγήσει με βάση το σχέδιο της οδηγίας αμέσως να διαβιβαστεί αυτή η περίπτωση στην ΕΠΠΟ. Αν υποθέσουμε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ανάγκη να έρθουμε σε επαφή με το Ηνωμένο Βασίλειο, τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου μια και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται εκτό πλαισίου ΙΠΠΟ, τότε θα μπορούσε η Eurojust ίσως ε, να διασφάλιζε τον συντονισμό μεταξύ των δύο κρατών ΙΠΠΟ ερχόμενη σε επαφή και συντονιστική τέτοια δραστηριότητα με ένα κράτος εκτός ΙΠΠΟ. Θα έπρεπε λοιπόν με αυτή τη δυνατότητα από πλευράς Παναμά ή Ελβετίας να μπορέσουμε άμεσα να διεκδικήσουμε ανάκτηση και θα πρέπει με τέτοιου είδους ε, συντονιστική δράση με κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσουμε, να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσω συζήτησης ε, και διακριβώσεων όταν διαπιστώνεται ότι τέτοιες περιπτώσεις ε, απατών οδηγούν σε φοροδιαφυγή υπονόμευση συμφερόντων Ευρωπαϊκής Ένωσης και συναποτελούν τότε ε, στοιχειώνουν, στοιχειοθετούν με συγχωρείτε περίπτωση παραβίασης ε, ευρωπαϊκής ε, νομοθεσίας τότε με το αντίστοιχο άρθρο υποχρεούνται τα κράτη-μέλη έναντι της Eurojust να δραστηριοποιηθούν ώστε μέσω για παράδειγμα του αντίστοιχου άρθρου να υπάρχει η δυνατότητα να διακριβωθεί ότι π.χ. μια άλλη εταιρεία, μια εταιρεία πορτογαλική μπορεί και εκείνη να συναποτελεί μέρος ενός πλαισίου φοροδιαφυγής που και πάλι οδηγεί σε υπονόμευση συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει αμέσως υποβολή στοιχείων για αυτή την περίπτωση στο EPPO. Αυτά βρίσκονται στην αρχική φάση αναφοράς αυτών των στοιχείων και περιπτώσεων και διαβίβασής τους. Μπορούμε να συνεχίσουμε και να δώσουμε περαιτέρω τέτοιες περιπτώσεις όπου πολλές άλλες χώρες εμπλέκονται και βρισκόμαστε και σε ένα πλαίσιο με συμμετοχή κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που μπορούν όλα αυτά να συσσωρεύουν ένα ποσό ε, κάποιων εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε λοιπόν θα πρέπει να μπορέσουμε να διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο σε αυτές τις διάφορες ε, πτυχές ε, ακόμα και στο ξέπλυμα χρήματος και βλέπουμε ότι τα θέματα δεν είναι μόνο δικαστικά αλλά και απόδειξης και τεκμηρίων σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος. Υποθέτοντας σε μια τέτοια περίπτωση ότι η Ολλανδία μπορεί να ε, έχει ρόλο, ε, ας το πω έτσι, κύριο ρόλο σε μια τέτοια ε, δραστηριότητα ως κράτος μέλος του ΕΠΠΟ, Ε, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν μια τέτοια περίπτωση να μπορέσει να δραστηριοποιήσει σε σχέση με την Ολλανδία και την ε, ίδια την δίωξη εκεί. Και έτσι δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος ότι άλλες ε, χώρες ε, θα μπορούν να ας το πω έτσι, υπεκφύγουν. Η ίδια η Ολλανδία θα μπορέσει να δράσει αποτελεσματικά. Εκεί λοιπόν αν υποθέσουμε τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο και βλέπουμε ότι πολλές δραστηριότητες ε, ε, βρίσκονται μέσα στο, στα πλαίσια του Ηνωμένου Βασιλείου, θα πρέπει σε σχέση με τις ε, ανακρίσεις και τη δίωξη να δούμε ότι ίσως θα μπορούσε να ζητηθεί από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να δεχθούν ότι η Ολλανδία θα είχε ε, καλύτερες δυνατότητες εκείνη να ασκήσει δίωξη. Βλέπουμε ότι μπορούν έτσι να διαφοροποιηθούν τα πράγματα, μπορούμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτόν τον κατάλογο που ε, μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω για το τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τη δίωξη εγκλημάτων εις βάρος ε, των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αναλαμβάνονται οι αναγκαίες δράσεις ώστε να μπορεί κανείς να ζητεί από τους, ε, τις αρμόδιες αρχές του πιο κατάλληλου κράτους να ασκήσουν τη δίωξη. Και βλέπουμε εδώ ότι και άλλες χώρες μπορούν να διαδραματίσουν ένα συγκεκριμένο ρόλο σε μια άλλη φάση για παράδειγμα Ιταλία, Δανία σε σχέση με τα έσοδα όταν υπήρχε τέτοια περίπτωση απάτης με θέματα μεταφοράς από την Δανία προς την Ιταλία μεταφοράς αγαθών και όταν ε, είχαμε και την περίπτωση σύλληψης ε, των αρμοδίων είναι αναγκαίο να υπάρξει ακριβής υπολογισμός ε, ώστε να δούμε ποια ακριβώς, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να υπολογιστεί μέρος της ποινής που καταλογίστηκε που επευλήθη ποιο τμήμα αυτής της ποινή ε, καλύφθηκε σε ε, κρατητήρια ή φυλακές της Δανίας ε, για τον συνυπολογισμό της, της πλήρους καταδίκης για το υπόλοιπο, για παράδειγμα στην Ιταλία. Και σε τέτοιου είδους περιπτώσεις σύγκρουσης δικαστικών θεμάτων υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε τέτοια κέντρα, κομβικά κέντρα συντονισμού. Το μήνυμα είναι που πρέπει να περάσει ότι ό,τι και να γίνει πρέπει να γίνεται εκ παραλίλου με τις δραστηριότητες ε, της Eurojust ώστε να διατίθενται τα κονδύλια με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ώστε να μπορούμε να ε, κάνουμε την πιο κερδοφόρα εποφελή χρήση και της πραγματογνωμοσύνης και του δυναμικού και των κονδυλίων μέσα στο πλαίσιο ακριβώς ε, αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Uh, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Νταν. Ε, Ευχαριστώ. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις ακούσαμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, το ξέρω. Κύριε Κούτς, τι μπορούμε να κάνουμε με τις περιπτώσεις ε, εγκατάλειψης δικών. Άκουσα ότι πολλές ε, υποθέσεις δεν προσάγονται καν στα δικαστήρια. Τι μπορεί να κάνει το δικαστήριο, να, η Επιτροπή ΚΡΙΜ να συστήσει, ε, η έκθεση για κολλήνο την οποία επεξεργαζόμαστε, κάτι που μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να μην σπαταλούμε και χρόνο και πόρους με αυτό το σοκαριστικό τρόπο. Κύριε Λιγκέτη. Μπορείτε να μας πείτε λιγάκι κάτι για τις κοινέ ερευνητικέ ομάδες. Η κυρία Επίτροπος, η κυρία Ρέντινγκ, νομίζω, αλλά άκουσα με τόσες ομιλίες που ξέχασα, μίλησε για 33, 33 κοινέ ερευνητικέ ομάδες πέρυσι. Μου φαίνεται μικρό το νούμερο αυτό. Γιατί? Γιατί είναι πολύ δύσκολο, είναι ακριβό αυτό το μέσο, αργό. Γιατί σίγουρα υπάρχουν πάνω από 33 διασυνοριακά εγκλήματα. Το νούμερο είναι σωστό, είναι λάθος. Αυτές οι κοινέ ομάδες είναι καλό εργαλείο, είναι επαχθές, διακρατικό μέσο, δεν δουλεύει. Είναι το μόνο που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Πέστε μου λίγα παραπάνω για αυτό το θέμα. Η τελική παρατήρηση, πολύ ενδιαφέρουσα, πολλά πράγματα ε, δεν υπάρχει πουθενά κάτι αντίστοιχο στην Ασία, στην Ινδία. Και εγώ είμαι στην αντιπροσωπεία με την Ινδία. Είναι απίστευτη ιστορία. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν έχει ε, αρμοδιότητε, δεν έχει ευθύνη για την καταπολέμηση του εγκλήματο. Ε, η Ινδία χρειάζεται ένα δικό τη ε, India Just, α πούμε. Δεν το έχουν σκεφτεί ακόμα. Ευτυχώ που εμεί το σκεφτήκαμε. Είμαστε μπροστά από όλου. Μπράβο μα. Δεύτερο ερώτημα οι, ε, οι σημαίες που μας δείξατε εκεί, η διαφάνεια με τις σημαίες, δεν είδα καθόλου την ελβετική σημαία. Συνεργάζεστε με, τη με την ε, Ελβετία. Άλλη ερώτηση. Μας ε, αναφέρατε το άρθρο 86. Ε, έρευνα, δίωξη, εκδίκαση. Ποιος κάνει τη δουλειά επί τόπου. Ποιος ψάχνει τα στοιχεία με το μεγεθυντικό φακό. Ποιος συλλαμβάνει τους εγκληματίες. Όχι εσείς βέβαια. Ούτε η Europol. Δεν μπορεί να το κάνετε αυτοί. Οι κοινέ ερευνητικέ ομάδε. Αυτή η δύσκολη συντονιστική προσπάθεια, α, πηγαίνετε να ελέγξετε αυτό το αυτοκίνητο κτλ. Έτσι γίνεται. Μου φαίνεται ότι κάτι χάνουμε εδώ πέρα, κάποιο κενό ή διαφωνείτε με αυτό το συμπέρασμα, αυτή η διαπίστωση. Ευχαριστώ κύριε Ντάν. Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που ήθελε το λόγο, ο κύριος Αγγιλάρ. Thank you. We're coming close to the final. Φτάνουμε στην τελευταία φάση της ακρόασης μια ερώτηση που είναι περίπλοκη. For a, summarized... Αλλά μπορεί να συνοψίσει όλη αυτή η συζήτηση από την εμπειρία που έχουμε. Που έχετε εσείς, ε, κυρία Κάνιν ως επικεφαλής ε, του Eurojust. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το στόχο του άρθρου 86 χρησιμοποιώντας την εμπειρία του Eurojust. Και έτσι να θέσουμε τις βάσεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με βάση την εμπειρία σας. Πόσες δυσκολίες συνδέονται και οφείλονται στις διαφορές των εθνικών νομοθεσιών. Παίζουν κάποιο ρόλο, δημιουργούν τα εμπόδια στη συνεργασία. Δημιουργούν προβλήματα στην δικαστική συνεργασία. Οι Ευρωπαίοι νομοθέτε που ασχολούνται με θέματα ποινική δικαιοσύνη μπορούν να κάνουν κάτι ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε από κοινού το σοβαρό διασυνοριακό έγκλημα. Ε, Ευχαριστώ κύριε Αγγιλάρ. Ο κύριος Ιακολίνο, τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που δεν άκουσα τις πρώτες παρεμβάσεις, τις πρώτες δύο παρεμβάσεις. Άκουσα μόνο την, κυρία, την τελευταία κυρία, την πρόεδρο του Eurojust. την κυρία Κόνιγκς. Έχετε 11 χρόνια εμπειρία από το Eurojust. Μεγαλύτερο συντονισμό τώρα, χάρη στο Eurojust, που προκύπτει από τα όσα είπατε με τα κράτη-μέλη. Πριν από καμιά ώρα, μια μισή ώρα, ακούσαμε την κυρία Ρέντινγκ. Δεν μας έδωσε πλήρες πληροφορίες ούτε για το χρονοδιάγραμμα, ούτε για τις προθεσμίες, μας είπε ότι έχουμε προχωρήσει απλώς στη σύνταξη του κειμένου για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και είπε ότι το Eurojust θα πρέπει να ξαναδεί ποιες αρμοδιότητες θα έχει. Ποιος, ποιος θα γίνει ανάμεσα σε αυτή την καινούργια ας πούμε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Όλαφ και την Eurojust. Εμείς πιστεύουμε ότι η Eurojust είναι μια κληρονομιά πληροφοριών που πρέπει να διατηρηθεί πολύ σημαντική. Εσείς, με βάση αυτή την εμπειρία, τι πιστεύετε. Μας μιλήσατε για τις μελλοντικέ δραστηριότητε δραστηριότητες που θα μπορούσε να έχει η Eurojust. Τι πιστεύετε για τις δραστηριότητε και τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πώς μπορούν να συνεπάρξουν αυτοί οι φορείς, αυτοί οι σημαντικοί οργανισμοί. Ούτω ή θα δούμε την πρόταση τη Κομισιόν, θα τη συζητήσουμε, θα την αξιολογήσουμε, θα υπάρξουν προφανώ τροπολογίε από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά σε τι γνώμη έχετε για αυτά. Πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Ο κύριος ο πρώτος ομιλητής, ο κύριος Κούλ, παίρνει το λόγο. Yes. <clears throat> Thank you very much. With respect to the... Uh, Σε σχέση με τις ε, επεξηγήσεις αυτές για τους πολύ υψηλούς ε, δείκτες ε, αποπομπής υποθέσεων, είναι πολύ δύσκολο να δοθεί μια απλή απάντηση γιατί είναι πολλοί οι λόγοι πολύ και ποικίλη. Όπως ξέρετε, αναλαμβάνουμε και διοικητικές διερευνήσεις με βάση τις ε, διοικητικές ε, διερευνήσεις και ανακρίσεις. Ακολουθούμε συγκεκριμένους ε, κανόνες και πολλές φορές η ίδια διερεύνηση γίνεται δύο φορές Δηλαδή γίνεται από διοικητικής πλευράς και ως προς το ποινικό σκέλος. Και αυτό καθυστερεί την όλη διαδικασία, είναι πηγή καθυστέρησης. Άρα πολλές υποθέσεις είναι σχηνοτενείς. Και γι' αυτό υπάρχει και υψηλό ποσοστό απόποντης. Και η κυρία Λιγκέτη πολύ σωστά είπε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ε, πολυσχηδείς καταστάσεις σε σχέση με το παραδεκτό αποδεικτικών στοιχείων. Ιδιαίτερα όταν τα αποδεικτικά στοιχεία συλλέγονται σε διεθνικό επίπεδο. Και γι' αυτό ορισμένες υποθέσεις ε, δεν μπορούν να προωθηθούν διότι λείπουν αποδεικτικά στοιχεία. Ε, πρόκειται για ιδιαίτερα επαχθείς διαδικασίες οι οποίες δεν μπορούν να φτάσουν σε αίσιο πέρας. Γι' αυτό χρειάζεται μία ενιαία Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή που και στη φάση δίωξης ανάκρισης να διέπεται από ένα ενιαίο πλαίσιο. Αυτό θα ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα εμπρός και ακριβώς αυτό είπαμε και στην παρουσίασή μας. Τώρα ως προς το μελλοντικό ρόλο της Όλαφ στα πλαίσια της συνεργασίας με την ΕΠΟ. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι αν συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, τότε ο ρόλος της Όλαφ θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, διότι δεν έχει νόημα ε, αυτές οι ποινικέ διαδικασίες να υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πρέπει να περάσουμε και από το διοικητικό πλαίσιο και μετά να διενεργηθούν έρευνες ως προς την ποινική ευθύνη. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα προαπαιτούμενα της διερεύνησης και να σταθούμε στο ποινικό σκέλος. Και αυτό σημαίνει ότι έτσι έχουμε λιγότερες υποθέσεις προς διερεύνηση από την Όλαφ και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους της Όλαφ στο μέλλον διαφορετικά. Δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε προσθέτοντας άλλον ένα παίκτη στο ευρωπαϊκό σκηνικό θα πρέπει να φτάσουμε σε οικονομίες κλίμακας και με ταχύτερο ρυθμό του παρόντος. Αυτή είναι και η πρώτη απάντηση στην ερώτησή σας. Ευχαριστούμε κύριε Κούλ. Η κυρία Λιγκέτη. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις για τις ε, κοινέ ερευνητικές ομάδες. Δεν έχω κοιτάξει τα στατιστικά στοιχεία ως προς τις JIT, ε, τις κοινέ ερευνητικές ομάδες. Ίσως ο αριθμός σας να είναι ακριβής. Γιατί χρησιμοποιήσαμε τόσο λίγο τις κοινέ ερευνητικές ομάδες. Εσείς επικαλεστήκατε αρκετούς λόγους, είναι δύσκολο να συσταθούν. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σύστασης των JIT των κοινών ερευνητικών ομάδων και θα πρέπει να υπάρχει μια πρωταρχική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών μελών του, των κανόνων του πώς θα λειτουργήσουν και ούτω καθεξής. Ακόμα και το νομικό πλαίσιο που ισχύει μας λέει ότι εάν αυτές οι κοινέ ερευνητικές ομάδες περάσουν από μία χώρα στην άλλη, αλλάζει ο ισχύον νόμος. Και αυτό δυσχεραίνει τα πράγματα ως προς την ε, κοινή διερεύνηση. Και ένα συγκεκριμένο κράτος ε, δεν μπορεί να συνεργαστεί με το κράτος Α με το κράτος Β, γιατί το νομικό πλαίσιο ή το νομικό περιβάλλον είναι διαφορετικό. Γι' αυτό είναι δύσκολο να έχουμε περισσότερες κοινέ ερευνητικές ομάδες. Αλλά υπάρχουν και πολλές ιστορίες επιτυχίας και η κυρία Κόνιγκς ίσως μπορεί να μας πει περισσότερα, γιατί και η Eurojust ε, συμμετέχει στα JIT. Ένα άλλο μείζον στοιχείο είναι ότι και στην κοινή ερευνητική ομάδα θέλουμε να συλλέξουμε αποδεικτικά στοιχεία τα οποία μπορούν να αχθούν ενώπιον του δικαστηρίου. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, αν ο νόμος να μπορέσουμε να συλλέξουμε αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία. Και χρειαζόμαστε ενιαίες εξουσίες για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Ίσως είναι δελεαστικό να πούμε ότι οι εκπρόσωποι της Εισαγγελικής Αρχής μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εθνικό δίκαιο. Έτσι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα μπορούσε να γίνει ευκολότερα αποδεκτή από πολιτικής άποψης και οι εκπρόσωποι της EPPO χρησιμοποιούν μια άλλη συνιστόσα εξουσιών από την Ευρωπαϊκή. Ίσως φαίνεται λειτουργεί σαν outsider η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Όμως με τις εθνικές αυτές εξουσίες θα φτάσουμε σε μπαλώματα και όχι σε μία ενιαία Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Και θα είναι πολύ ε, δύσκολο να ορίσουμε αυτή την εισαγγελική αρχή με πραγματικές διοκτικές εξουσίες. Έχουμε λίγα λεπτά για να μας απαντήσει η κυρία Κόνιξ. Madam Chair. I uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για αυτά τα λίγα λεπτά με τις έξι ερωτήσεις θα είμαι σύντομη στην απάντηση. Ναι, υπάρχει δικαστική συμφωνία για την δικαστική συνεργασία με την Ελβετία. Πέρυσι άρχισε να ισχύει αυτή η συμφωνία. Οι σημαίες που είδατε στην οθόνη οφείλονται στους ε, δικαστικούς ε, που οδήγησαν η Eurojust να εργάζεται μέσα σε ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο, διότι έχουμε και την, ε, την σύνδεση αυτή με τα ε, υπόλοιπα κράτη. Έχουμε και με την, ε, τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Νορβηγία και την Κροατία. Έχουμε την Ελβετία που έχει κιόλας ε, εντυπωσιακές επιδόσεις ε, σε διασύνδεση με τη Eurojust ε, στο κοινό έργο. Και σε σχέση με τους δικαστές αυτούς θα έλεγα ότι είναι αποτελεί η δυνατότητα αυτή μια εικόνα των επιτευγμάτων που έχουμε επιτύχει. Τώρα, σε σχέση με τις διακριβώσεις ε, ε, και τις διοκτικές δράσεις για την προσαγωγή των υπευθύνων ποινικά στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη ε, πείρα. Όμως έχοντας ευήκονους με το οποίο παρακολουθήσαμε δηλώσεις και τοποθετήσεις άλλων και από πλευράς ε, της Επιτροπής ε, αυτό που υποθέτουμε είναι ότι θα είχαμε ένα ας το πω έτσι, μια δράση μέσα στο EPPO με την συντονιστική δράση και των εισαγγελέων από πλευρά κρατών μελών για την παρακολούθηση αυτών των περιπτώσεων για την προσαγωγή των υπεύθυνων στα δικαστήρια, στη δικαιοσύνη, με την ροή των πληροφοριών και ανταλλαγή πληροφοριών από και προς την ΕΠΠΟ. Έχουμε ήδη ένα σύστημα για τη ροή αυτών των πληροφοριών με την Eurojust που μπορεί να διαθρώνεται δομικά και στα ίδια τα κράτη-μέλη και μέσω των εθνικών συντονιστικών συστημάτων της Eurojust με άμεσες επαφές με τις, ε, τους εθνικά υπεύθυνους ε, από πλευράς Eurojust ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και την δίωξη ώστε μέσω αυτού του πλαισίου να διασφαλίζεται η δομημένη διαθρωμένη δράση και να υπάρχει μια αποτελεσματική διασύνδεση. Αυτό θα πρέπει να γίνει και στο μέλλον, δοθεί συνέχεια σε αυτή την συνιστόσα να διαπιστωθούν οι δυνατότητες ε, λειτουργίας ε, ενός συστήματος που θα προσαρμόζεται στις ε, εξειδικευμένες ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με την δυνατότητα να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Αυτό είναι εκείνο το οποίο μελλοντικά σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε με τις ανακρίσεις και διακριβωτικές δράσεις προσαγωγή των υπεύθυνων στη δικαιοσύνη, σημαντική διασύνδεση που εξασφαλίζεται με τους αρμοδίους των κρατών μελών έτσι. Για την ερώτηση που έγινε από πλευράς του κυρίου Προέδρου Λόπες Αγγιλάρ, από πλευράς Eurojust έχουμε 30 διαφορετικά συστήματα, 23 διαφορετικές γλώσσες και παρόλα αυτά καταφέραμε να συντονίσουμε και να συντονιστούμε και να διευκολύνουμε το έργο αυτό ώστε να μπορέσουν οι ύποπτοι να προσαχθούν στα δικαστήρια και να δικαστούν. Έχοντας παρακολουθήσει τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει αναλυφθεί πρωτοβουλία και δράση ώστε να υπάρχει ένα σχέδιο οδηγίας για την δίωξη και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ανάγκη που υπάρχει και πρέπει να καλύψουμε. Έχουμε και την ανάγκη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων. Υπάρχει απουσία στατιστικών στοιχείων. Επειδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει από πλευρά ορισμών, δεν καλύπτεται επαρκώς από πλευρά ορισμού η πτυχή αυτή. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένε ποινικέ διαδικασίε όσον αφορά το δικονομικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με τον πιο σωστό τρόπο. Να μπορεί ο ένας να συντονίζεται με τον άλλο και επανερχόμενοι στην διευρυμένη συνεργασία έχουμε και πιο περίπλοκες καταστάσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με βάση τους κανόνες ε, μεταξύ των ε, νομικών συστημάτων και με βάση τις διάφορες ε, συμβάσεις και άλλους εξειδικευμένους κανόνες και διατάξεις. Ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη, με άλλα λόγια, για την διασφάλιση των σωστών συντονιστικών δράσεων. Όλα αυτά πρέπει να είναι εφικτά και να μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Και από πλευράς Eurojust και Europol τονίστηκαν αυτές οι πτυχές ήδη για τον ρόλο της ε, Eurojust ε, π.χ. και για τον, την Όλαφ που το, η Όλαφ διασφαλίζει το τεχνικό επίπεδο ε, ερευνών μέσω της μονάδας της και έχει και την τεχνική πραγματογνωμοσύνη. Η Europol είναι η ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αστυνομικής και Δικαστικής Συνεργασίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε τον στόχο όλες αυτές οι προσπάθειες να συγκλίνουν προς μια κοινή κατεύθυνση σε ένα κοινό πλαίσιο. Τα διάφορα, διαφορετικά πρότυπα τώρα τα οποία βρίσκονται υπό εξέταση δεν μπορούμε να προδικάσουμε τι ακριβώς θα γίνει και ποιο πρότυπο θα υιοθετηθεί αλλά Eurojust θα πρέπει μέσα στο πλαίσιο του EPPO να οριμάσει, να οδηγήσει τα πράγματα αυτά να οριμάσουν και μέσω του άρθρου για παράδειγμα 6 να διασφαλιστεί μια ξεχωριστή μονάδα με ξεχωριστές αρμοδιότητες όσον αφορά το άρθρο 86 και να μπορέσουμε έτσι να δραχθούμε των ευκαιριών των κονδυλίων της Eurojust με βάση τις προηγούμενες, ε, την προηγούμενη πείρα και πραγματογνωμοσύνη που έχει συλλέξει η Eurojust. Το ίδιο ισχύει και για την πραγματογνωμοσύνη από πλευράς ε, της Europol και της ε, Olaf. Τα ίδια πρέπει να ισχύουν. Και έτσι μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτά είναι τα σχέδια που έχουμε ενώπιόν μας και μπορούν να προχωρήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κόνιξ. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες, τους συναδέλφους για την ακρόαση. Έχετε όλες τις πληροφορίες ως συνήθως και τις εκθέσεις στη διάθεσή σας. στο site της Επιτροπής μας.